Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκε να περιμένετε. Ε, ζητώ ιδιαίτερο συγγνώμη από τον κύριο Άγνιο που διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση, αλλά σκέφτηκα επειδή είναι σήμερα Δευτέρα και σήμερα φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάδελφοι να αφήσω λίγο περισσότερο χρόνο. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη, αγαπητοί συνάδελφοι. Το σημείο 6, παρουσίαση δηλαδή του σχεδίου γνωμοδότησης για το ελαιόλαδο, αναβάλλεται για την συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου, ύστερα από αίτημα του συντάκτη της γνωμοδότησης. Οπότε η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στη μία πολύ λίγο χρόνο μένει δηλαδή για τι προθεσμίε. Επίση, ε, αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και έχουμε συνεδρίαση σε 16 γλώσσε, λέει ο πρόεδρο, 15 κανονικά. Ε, έχετε λάβει και το διορθωτικό μια νομοθετική πράξη. Η γραμματεία σα μοίρασε και μάλιστα σε όλε τι μεταφράσει ε, το διορθωτικό για τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις. Δηλαδή, τον κανονισμό 1306 του 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινή γεωργικής πολιτικής που καταργεί άλλους κανονισμούς. Το πρόβλημα είναι στο ότι οι συνάδελφοι μας εκπρόσωποι ε, από τη Διεύθυνση Νομοθετικών Πράξεων ε, εξέτασαν το διορθωτικό, μας ενημέρωσαν ότι ε, έχει συμφωνηθεί από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπάρχει μάλιστα μία σημείωση διορθωτική στη σελίδα 603 που έχει αμυγός τεχνικό χαρακτήρα, αφορά ένα τελείως τεχνικό ζήτημα, οπότε με βάση το άρθρο 231 το διορθωτικό θα πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια μετά από εξέταση που θα γίνει στην αρμόδια Επιτροπή. Οπότε, αν δεν υποβληθούν ενστάσει ή παρατηρήσει μέχρι το πέρα τη συνεδρίαση για το διορθωτικό αυτό, θα προτείνω ε, να το διαβάσουμε λέγοντα ότι ομόφωνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή μα. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις να εγκρίνουμε τα πρακτικά τη συνεδρίαση τη 25η Σεπτεμβρίου. Αν μέχρι το πέρα συνεδρία δεν υποβληθούν παρατηρήσει, θα θεωρηθούν και αυτά ω εγκεκριμένα. Περνάμε στο σημείο 4. Την γνωμοδότηση για τον κανονισμό Omnibus. Ασχολεί, ασχολούνται με το θέμα αυτό οι κύριοι Ντές και Ντεκάστρο, όπως ξέρετε. Ε, πρώτα ο κύριος Ντεκάστρο, τώρα ο κύριος Ντές και μας, θα μας ενημερώσει ο κύριος Ντές για τις εξελίξεις των συζητήσεων με το Συμβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ θετικές οι διαπραγματεύσεις, στέφθηκα με επιτυχία και θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή μας αλλά και την Προεδρεύουσα το Συμβούλιο χώρα για τις πολύ επικοδομητικές συζητήσεις που κατέληξαν, όπως σας είπα, σε αίσιο πέρας, παρά τα δύσκολα προβλήματα και τις δύσκολες συνθήκες. Κατόρθωσαν πάντως τα θεσμικά όργανα να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία. Ε, ο κύριος Δεκάστρο επίσης συμμετείχε στη διαδικασία και διευκόλυνε τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Και βοήθησε και τον κύριο Ντές, ε, μια και ήταν ο προκάτοχός του στα θέματα αυτά. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις πάντως, α, ακαθόδες. Αλλά θα μας ενημερώσει για όλα αυτά ο αρμόδιος συντάκτης γνωμοδότης, ο κύριος Άλμπερ Ντές. Παρακαλώ κύριε Ντές. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου επεκτείνοντάς τις ταυτόχρονα στους ε, συναδέλφους από τις άλλες επτά ομάδες που είχαν τα ίδια θέματα στι αρμοδιότητες τους και τη συμμετοχή βέβαια στον τριμερή διάλογο και οι οποίοι έχουν επισημάνει ότι συμφωνούν με το τελικό αποτέλεσμα και το στόχο τον οποίο επιτύχαμε. Ήταν ε, πολύ καλές οι διαπραγματεύσεις. Καταλήξαμε όμως σε κάτι που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο στην πολιτική, από ένα σημείο αφετηρία, σημεία αφετηρίας αρκετά διαφορετικά, να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Και ευχαριστώ όλους τους ε, συνεργαστέντες, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και, το, και του Πάολο, ο οποίος έκανε δυτικές προσπάθειες, όπως και την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το πολύ καλό κλίμα των διαπραγματεύσεων. Ξεκινήσαμε με διαφορετικές θέσεις και επόψεις, αλλά φτάσαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Και θέλω να ενημερώσω για τα περαιτέρω και το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Γκρέσλε, γιατί προχωρεί αυτό ανεξάρτητα από την υπόλοιπη διαδικασία, είχε πει η κυρία Γκρέσλε λοιπόν ότι θα ε, παρακολουθήσει το θέμα, αλλά πρέπει μέχρι την Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα, στο Προεδρείο να έχουμε λάβει απόφαση εάν θέλουμε μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2018 να είμαστε σε θέση να έχουμε τη θέση εφαρμογή του νέου κανονισμού και πρέπει ναι, να είμαστε σε θέση να θέσουμε σε εφαρμογή τις ε, τροπολογίες. Ιδάλλως πάμε για το 2019 και έχουμε χάσει ουσιαστικά ε, ολόκληρη, έχουμε, έχει μείνει μόνο το τέλος αυτής της ε, περίοδου της γεωργικής. Άρα πέμπτη της επόμενης εβδομάδας στο Προεδρείο πρέπει να ληφθεί απόφαση για να είμαστε για τις 30 ε, ενδεκάτου εδώ στις Βρυξέλλες στη Μήνη Ολομέλεια έτοιμη για την ψηφοφορία 22 βέβαια στην Επιτροπή μας, 22 11 θα πρέπει να γίνει στην Επιτροπή Γεωργίας η ψηφοφορία και όπως είπα Προεδρείο, πρέπει να λάβει απόφαση το Προεδρείο την επόμενη Πέμπτη για να ε, προχωρήσει το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, ε, για τα επιμέρους σημεία. Κυρία, ε, συγκεκριμένα προβλήματα, μεγάλα προβλήματα δεν είχαμε για τον οριζόντιο κανονισμό. Για τους επιμέρους κανονισμούς πάνω απ' όλα ήταν σημαντικοί οι ορισμοί που έχουν να κάνουν με την διαρκή πράσινη έκταση. Εδώ είδαμε ότι θα είχαμε σημαντικές δυσκολίες, αλλά δεν θέλησε κανείς να επιμένει έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και σε σχέση με το περιβάλλον και βεβαίω καταλήξαμε σε μια λογική, ορθολογική, συμβαστική λύση που πιστεύω ότι θα προχωρήσει με ακόμη πιο λογικές λύσεις την προσεχή μεταρρύθμιση της ΚΑΠ γιατί θα ήταν αντιπαραγωγικό να μην έχουμε τους κατάλληλους ορισμούς Επτά χρόνια η διατήρηση της πράσινης έκτασης είναι μια λύση λογική και εφικτή. Αλλά θα ήταν καλύτερο να έχουμε τη δυνατότητα για τα πέντε χρόνια. Επίσης, οι μειονεκτικές περιοχές, διαφορετικοί ορισμοί και οι θεωρίες των κρατών μελών. Από το 2018 στον, ε, προχωρούν τα κρατημέλη στην εγκατάλειψη του αρνητικού καταλόγου έρεται ο περιορισμός στην έκταση ανεκτάριο, δηλαδή εφόσον υπάρχει πράσινη ε, έκταση, ορίζει την ε, απαγόρευση της χρήσης ε, φυτοπροστατευτικών ουσιών με της πράξη ο Επίτροπος. Μετά έχουμε το Έχουμε διάφορα σιτηρά τα οποία εξαιρούνται και βέβαια μετά το ταξίδι μας στην Κροατία συζητήσαμε διάφορα θέματα. Έχουμε στην ανάπτυξη της υπαίθρου προτείνει τις λύσεις για, και για την κοινή οργάνωση της αγοράς και εκεί έχουμε επιτύχει με τη συνεργασία των συναδέλφων διαφορές ε, ε, προόδους και γενικά πιστεύω ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα καλό για την ΚΑΠ και το σημαντικό πλέον είναι να τεθεί εγκαίρως σε εφαρμογή η νέα πρόταση. Νομίζω ότι μπορούμε με τη Γαλλία και τη Γερμανία να έχουμε καλά αποτελέσματα. Θα προσπαθήσει και η Γκέμποργκ Κρέτσλε προς την κατεύθυνση αυτή και με τον τριμερή διάλογο βέβαια πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα ώστε να προχωρήσουμε στην ε, ε, ολοκλήρωση διαδικασίας για το splitting. Αυτά από πλευρά μου και βέβαια θα πρέπει να ακούσουμε και τον κύριο Δεκάστρο, Λέω, ο Πρόεδρος. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω και εγώ δύο λόγια. Θα συμφωνήσω με τον Αλμπερντές, εξαιρετική δουλειά και η συνεργασία. Η Επιτροπή μας νομίζω μπορεί να είναι υπερήφανη για τη δουλειά που έγινε. Κάναμε όλη τη δουλειά και στις 12 Οκτωβρίου καταλήξαμε σε μια συμφωνία που σε όρους όχι μόνο ουσίας περιεχομένου, που λίγο πολύ ε, προεξόφλησε και ο Αλμπερντές, αλλά και σε όρους χρόνου, γιατί καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ταχύτατα σε χρόνους δηλαδή που μας επιτρέπουν να θέσουμε σε εκκίνηση μια διαδικασία την διαδικασία για την αποκοπή, το splitting από το υπόλοιπο του κανονισμού Omnibus και να επιταχύνουμε τη θέση εφαρμογή έτσι ώστε από την 1η Ιανουαρίου του 2018 να έχουμε το σύνολο των κανόνων που αφορούν τη γεωργία από τον κανονισμό Omnibus σε εφαρμογή. Αν συμφωνεί ο κύριο Σικέρης και βέβαια και ο Φιλίπ από τη Γραμματεία της Επιτροπής θα μπορούσαν ε, να μας ετοιμάσουν μια πολύ σύντομη παρουσίαση των ε, προσεχών βημάτων γιατί ε, κάνουμε μια κούρσα εναντίον στο χρόνο αυτή τη στιγμή, εναντίον στο ρολόι. Όλα τα κεφάλαια του Omnibus έχουν παρουσιάσει καθυστερήσει, σημειώνω. Και ίσως το πιο σημαντικό τέλεχος που είναι ο προϋπολογισμός μπορεί να περάσει σε περίοδο μετά τους πρώτους μήνες του 2018 σε έγκριση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το splitting, ο διαχωρισμός δηλαδή και να κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε ώστε η τελική ψηφοφορία στη μήνυ ολομέλεια των Βρυξελών να επιτρέψει την δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα μέσα στις ε, χριστουγεννιάτικε διακοπέ ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κύριε Τεκάστρο. Ο κύριο Αντριέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε ικανοποιημένοι και από το έργο του κ. και από το έργο του προκατόχου του και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ειλικρινά ότι οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και το έργο των εκπροσώπων μας αξιέπαινο. Αλλά ας μην γελιόμαστε. Ε, θα πρέπει να δούμε πέραν των αλλαγών τι κρύβεται πίσω από τη στάση του Συμβουλίου. Γιατί ουσιαστικά θέλει να ιδιωτικοποιήσει την ΚΑΠ και να ε, απομακρύνει το, τη δέσμευση του δημοσίου ε, στην ΚΑΠ και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και να μας θορυβεί γιατί φαίνεται ότι θέλουμε να ε, οδηγηθούμε σε μια επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και όλο και μεγαλύτερη απομάκρυση της από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Κάτι τέτοιο όμως θα υπογράψει τη θανατική καταδίκη της ΚΑΠ. Μια επανεθνικοποίηση και απομάκρυση από το κοινοτικό χαρακτήρα. Επίσης, πολύ πιστεύουμε αδίκως ότι η δυσλειτουργία των αγορών και η αστάθεια που ε, ε, ε, επιτεχήθηκε από τις εμπορικές συμφωνίες πάσης φύσεως και το καταγγείλαμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να διορθωθούν μόνο με κάποιες μηχανισμούς διαβεβαίωσης. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο γιατί δεν συνάδει κάτι τέτοιο ούτε με τις δικές μας επιθυμίες. Και παρά τις ε, δεν θεωρώ ότι οι μηχανισμοί αυτοί αρκούν. Και αυτοί που θα βγουν κερδισμένοι από κάτι τέτοιο είναι μόνο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τη μεταφορά άμεσων ενισχύσεων προς τα ασφαλιστικά συστήματα γιατί όλοι θεωρούν ή προσπαθούν να μας πείσουν ότι στην ασφάλεια βρίσκεται ε, η λύση. Και θα πρέπει επίσης όλοι οι παραγωγοί να έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίσουν τις οδιές τους ε, και να καταβάλουν τα ασφάλιστρα. Δεν νομίζω ότι ε, οι ασφάλειες θα μα λύσουν όλα τα προβλήματα στο σύνολο του κλάδου. Επίση, η αλλαγή των κανόνων του ΠΟΕ που δίνει μεγαλύτερε ευθύνε στους επαγγελματίε, στην οργάνωση τη ε, επιστηστικής αλυσίδα, δίνοντα περισσότερα περιθώρια ω προ του κανόνες του ανταγωνισμού και αυτό εντοπίστηκε ε, και αναφέρθηκε και ευχαριστώ τον κύριο Νταντέν για τις προτάσεις του. Είναι απαραίτητο στάδιο, αλλά δεν νομίζω ότι αρκούν οι προτινόμενες αλλαγές για να επαναφέρουμε μια ισορροπία στην έλλειψη του διαπραγματευτικού της διαπραγματευτικής ισχύω ε, των παραγωγών και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Τίποτα δεν είχαμε για τη διαχείριση και πρόληψη των κρίσεων και μία ελάχιστη ρύθμιση αγορών, κάτι που είναι απαραίτητο ε, για την σταθερότητα των τιμών και την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος. Ούτε σήμερα βρισκόμαστε στο πυρόβλητο νέων κρίσεων. Γιατί είχαμε κρίσεις στο γαλακτοκομικό τομέα και δεν θα πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους αυτές οι κρίσεις και στις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Είπα το, και το επαναλαμβάνω, ευχαριστώ του συναδέλφου για το έργο του στον κανονισμό Omnibus, αλλά θα πρέπει να βρισκόμαστε σε, σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση και να μην γελιόμαστε, γιατί υπάρχουν πολλά προβληματικά σημεία που θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Ευχαριστώ, κύριο Νταντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ε, συμφωνήσω με τα σχόλια των συναδέλφων Τέσ και Δικάστρο. Και να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία της Επιτροπής ε, που μας ε, επικούρησε σε όλη αυτή την προσπάθεια και μας βοήθησε να προχωρήσουμε. Εδώ και πολλούς μήνες επανειλημμένος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφραζε τα επιχείρηματά του και προσπάθησε να ε, γίνει δεκτή η γνώμη του. Είχαμε τις εκθέσεις ε, Μαγκίνες και Ντελαέ και επιτέλους ε, εισακούστηκε η γνώμη μας και για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά το, την κοινή οργάνωση αγοράς, 39 από τις 53 τροπολογίες μας έγιναν δεκτές και καλύφθηκαν από τη διακήρυξη. Πάνω από τις 75% των τροπολογιών δηλαδή έγιναν δεκτές από εμά, κάτι που δείχνει ότι εργαστήκαμε συλλογικά πολύ καλά. Επίσης, ε, για τα απορροκυπευτικά. Τροποποίησαμε άρδιν την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής υπερημών, ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες δράσεις διαφοροποίησης και εδραίωσης των αγορών, το coaching και εθνική αρρωγή στις χώρες που έχουν κάποια σημεία για την ε, συλλογική οργάνωση, σε ό,τι αφορά τον ίνο τα αιτήματά μας ε, για την κάλυψη, για, την, για τις ονομασίες προέλευσης, για, την, για τον εμπλουτισμό, όλες μας οι προτάσεις έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τον Ινό. Σε ό,τι αφορά για τη σύναψη συμβάσεων, ε, ε, τον αθέμητο ανταγωνισμό και, την οργάνωση, Έχουμε το μεμονωμένο δικαίωμα για ατομική σύμβαση των γεωργών, επίση τη δυνατότητα διαπραγμάτευση ε, στο περιθώριο των συμβάσεων για ε, ρήτρε ε, επιμερισμού τη προστιθέμενη αξία σε περίπτωση που αυξηθεί η αξία από τη στιγμή τη υπογραφή τη σύμβαση και τη παράδοση του προϊόντος, όπως γίνεται στα ζαχαρότευτλα. Επίση, για του περιβαλλοντικού και υγειονομικού κινδύνου και τον επιμερισμό τη προσθέμενη αξία, επίση πέρασαν τα θέματα μα. Στήσαμε δήλωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάλυση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόταση κειμένου για το θέμα αυτό το 2018. Και τέλο, ένα πολύ επίσημα σημαντικό θέμα, την κατάργηση τη ε, οριστική προθεσμία για το πακέτο του γάλακτο που ήταν κανονικά το 2020. Τώρα πια δεν έχουμε τέτοια ημερομηνία καταληκτική για το γάλα. Πάντως, οι οργανώσεις παραγωγών και οι συνεταιρισμοί, οι γεωργικοί συνεταιρισμοί ε, βλέπουν τα προνόμια τους να αναγνωρίζονται πια στο κείμενο, γιατί προβλέπονται ρητά από τον κανονισμό, ότι υπάρχει, προβλέπεται εξαίρεση από το δίκαιο ανταγωνισμού για τις οργανώσεις αυτές, οργανώσεις παραγωγών και, συνε, και τις, ε, τους συνεταιρισμούς, ώστε όλοι οι τομείς παραγωγής μπορούν ε, να διαπραγματεύονται σύμβαση με κοινή σύμβαση και να ε, βελτιστοποιήσουν το κόστος της παραγωγής. Σε ό,τι αφορά το δίκαιο ανταγωνισμού, καταφέραμε να μπορούμε να α, ρωτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα συγκεκριμένο σχέδιο εμπίπτει στην εξαίρεση από το δίκαιο ανταγωνισμού και ε, επέκταση της δυνατότητας εξαίρεσης από το δίκαιο ανταγωνισμού σε περίοδο κρίσης για τις διαπαγγελματικέ οργανώσεις συνεταιρισμού ή όσου καλύπτονται από ε, ονομασίες προέλευση και επίσης χρήση ω έσχα της λύσης αυτού του μηχανισμού ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο κείμενο του 2013 ε, το, ο μηχανισμός αυτός ήταν μόνο η τελευταία λύση σε περίπτωση που ήταν αποτελεσματικέ όλε οι προηγούμενε. αλλά τώρα έχουμε βελτιώσει αυτό το θέμα. Επίσης, ε, Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουν και οι παραγωγοί αυτές, αυτή την πρόοδο θα έχουμε πραγματικά αυτά σημεία για να, και σημαντικά άρθρα για να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο του κ. Αντριώ για τις ασφάλειες, όντως είχαμε μεγάλες δυσκολίες στο να πείσουμε το Συμβούλιο να δεχτεί κάποια μέτρα για τη διαχείριση των κρίσεων και αυτό που επιτύχαμε ήταν ε, το ελάχιστο που απαιτούσαμε. Ε, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ενίσχυση, αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία στα κράτη-μέλη. Θέλουμε μια πολιτική διαχείριση των κρίσεων και όχι ετήσια. Και θέλουμε ένα πακτολό που θα διαμορφώνεται από τα πλεονέσματα κάθε χρονιάς και που θα επιστρέφεται ε, στα κράτη-μέλη μετά απο δυο δύο-τρία χρόνια αν, αν δεν εκταμιεύεται ή δεν απορροφάται το σύνολο των κονδύλων του πακέτου Επίσης, τα αμοιβαία κεφάλαια ουσιαστικά οι ασφάλειες ουσιαστικά προϋποθέτουν αποθέματα οικονομικά για τα οποία δεν έχουμε σήμερα κρατικούς μηχανισμούς που να επιτρέπουν τη σύσταση τέτοιων αποθεματικών. Και σήμερα που αντιμετωπίζουμε πολλές κρίσεις, όχι μόνο γεωργικές, αλλά και τη μεταναστευτική και την κρίση της ασφάλειας, το να προτείνουμε αιτήσια ε, ε, διόγκωση του προπολογισμού θα είναι και δύσκολη για να μην πω απίθανη. Αρκεί να μιλήσουμε με του συναδέλφου μα από την Επιτροπή Προπολογισμών για να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουμε τη συμφωνία τη ε, Επιτροπή Προπολογισμών για τα θέματα αυτά για να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον Άλμπερτ και τον Πάολο για την ε, δουλειά που έκαναν δύσκολη οπωσδήποτε δόθηκε μεγάλος αγώνας νομίζω ότι τελικά το θέμα είναι το αν βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο εγώ είμαι αισιόδοξο. νομίζω ότι πήραμε περισσότερα από ότι αρχικά αναμέναμε γι' αυτό και πραγματικά ε, θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους για τη δουλειά που έκαναν αλλά πρέπει να πω ότι ακόμα δεν έχω πιστεί για το ότι η ασφάλιση είναι ο καλύτερος ε, δρόμος για να στηρίξουμε τη Γεωργία. Ποτέ δεν είχα πιστεί και δεν έχω πιστεί ακόμα. Αλλά αυτό είναι. Δεν είναι της ε, στιγμής. Επίσης ε, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού φαίνεται ότι θα μας ακολουθεί από εδώ και μπρος ε, σε κάθε βήμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Και μου κάνει λίγο εντύπωση για το ότι δεν κάνει τίποτα για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που ελέγχουν την αγορά και υπαγορεύουν τις τιμές. Αν έκαναν τίποτα. Προς τα εκεί ε, θα ήμασταν και εμείς ε, κάπως πιο ε, ευέλικτοι, αλλά όταν δεν κάνουν την δουλειά τους σωστά δεν μπορώ και εγώ να είμαι ικανοποιημένος. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ εξ ονόματος της ΑΛΔΕ να ευχαριστήσω τον Άλμπερτ ε, και τον Πάολο και τους συνεργάτες και την γραμματεία. Απαιτήθηκαν πολλές ε, συναντήσεις ε, και διαπραγματεύσεις και το αποτέλεσμα αυτό μπορούμε να το δεχτούμε και εμείς ένας ευρύτατος συμβιβασμός. Για εμάς βεβαίως είναι σημαντικότερο το, σημαντικό το ότι έχουμε το splitting και ότι από 1η 2018 έχουμε απλοποιήσεις για τους αγρότες. Βεβαίως κάποιες δυσκολίες ε, έχει η ομάδα μου με τον ε, κοινό κανονισμό της αγοράς. Δεν το έχουμε κρύψει ποτέ και όταν διαβάζουμε και τον γερμανικό τύπο, ειδικά από την πλευρά των ε, συνεταιρισμών, βλέπουμε ότι είχαμε δίκιο στις αντιρρήσεις μας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε την ε, μεγάλη, την ευρύτερη εικόνα και τις βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει εδώ και πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον. Οπότε θα στηρίξουμε αυτήν την πρόταση και ελπίζω και στην ψηφοφορία να έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, οφείλω να πω, και δεν είχα συνειδητοποιήσει την σημασία απλών λέξεων όπως θα ή επιτρέπεται κτλ. Αλλά τελικά το αντιλήφθηκα γιατί Νομίζω πως έχουμε κάποια καλά νέα για την νέα γενιά αγροτών και την ανανέωση. Ε, και έτσι τώρα εάν ένα κράτος το θέλει μπορεί να επιτρέψει σε έναν αγρότη να μείνει ως νέος αγρότης για πέντε χρόνια ακόμα και αν ε, ήταν στο ίδιο καθεστώς και πέντε χρόνια πριν. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Και Ελπίζω να γίνει υποχρεωτικό αυτό, αλλά έχουμε μια κατάσταση όπου στη δική μου τη χώρα, παρά το ότι υπάρχουν εδώ σε αυτή την Επιτροπή Ιρλανδοί που λένε ότι θέλουν να κάνουν κάτι για το θέμα, δυστυχώς η δική μου η χώρα επέμεινε στο να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου μπορεί μια χώρα να μην δώσει λεφτά στους νέους αγρότες και δυστυχώς η δικιά μου η χώρα επέμεινε γι' αυτό. Ε, εγώ δεν τρέπω προσωπικά, αλλά αυτοί που το πρόθεσαν θα έπρεπε να ντρέπονται. Όπως είπαν κι άλλοι βεβαίως ε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, οπωσδήποτε δεν είναι καλά τα νέα με την ασφάλιση και την εισαγωγή χρηματοοικονομικών μέσων πάλι δίνει λεφτά ο αγρότης και αυτό δεν είναι καλό. Αλλά η κύρια απογοήτευσή μου, όπως σας είπα, είναι από τους συμπατριώτες μου. Τέλος πάντων, τι να πω, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ναι. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και τα μελλοντικά βήματα στη διαδικασία αυτή. Έγιναν κάποια πρώτα βήματα ή εκφράστηκαν κάποιες, κάποιοι φόβοι για τον επιμερισμό ε, των γεωργικών εκτάσεων. Ε, τελικά ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην γίνει αυτή η κατανομή, αλλά ε, Εμεί κάναμε ό,τι μπορούσαμε και το δικό μα ε, τμήμα προωθήθηκε. Οι καθυστερήσει γίνονται αλλού. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα. Αν θα μας επιτρέψουν να, να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η Γεωργία ήδη από τον επόμενο χρόνο θα μπορούσαν να έχουν πολλές διευκολύνσεις που μας τις παρουσίασε ο κύριος Δες. Οπότε θα μπορούσαμε από πολύ διαφορετική θέση να το διαπιστώσουμε και να είμαστε σε άλλη θέση εν και της χρονιάς των ευρωεκλογών του 2019. Θα δώσω το λόγο και στον επικεφαλής της γραμματείας για να μας ε, εξηγήσει τα διαδικαστικά. Αλλά θα ακούσουμε πρώτα και τους προσώπους των υπόλοιπων ομάδων και μετά θα δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Ντες για να απαντήσει. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα-δύο πράγματα μόνο που δεν προλαμβάνω νωρίτερα να επισημάνω. Ε, προς την ορθή κατεύθυνση βαίνουν μεν οι βουλήσεις όπως εκδήλωνονται, αλλά στην ουσία δεν βλέπουμε τίποτε το καλό, ούτε απλοποίηση, ό,τι και να λέμε, υπέρ του Γεωργού για την ΚΑΠ. Ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι πανταχού παρόν, είναι ακόμη παρόν. Και με όλη τη βούληση και το καταγγέλουμε πάντα με το συνάδελφο Φερό ότι δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία όσο συνεχίζουμε σε αυτή την πολιτική της παγκοσμιοποίησης. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Κύριε Ευρωβουλευτά, έγινε ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει και αυτό να το αναγνωρίσουμε και να το εκτιμήσουμε. Δεν είχαμε από την αρχή τόσο γρήγορο ρυθμό και τόσο καλή πρόοδο. Ευχαριστώ. Κύριος Γιάρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βεβαίω, να ρωτήσουμε τον καθέναν χωριστά από εμά εδώ στην Επιτροπή. Θα έχουμε και διαφορετικέ επιθυμίε και προτιμήσει, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το σύνολο. Και ήταν πάρα πολύ καλή ο συνολικό συμβασμό και πρέπει να συγχαρούμε του εισηγητέ. Και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Και θα έλεγα λίγο πολύ να δούμε και την ανταμοιβή αυτή τη αυστηρή τηρήση του χρονοδιαγράμματο, γιατί τηρήσαμε το λόγο μα, την υπόσχεσή μα, φέρουμε το αποτέλεσμα την ώρα που πρέπει. Ε, Α μην βρεθούν να τιμωρούνται εκείνοι που δεν πρέπει. Τηρήσαμε, όπω είπαμε, το λόγο μα. Για να μην πω ότι οι συγητέ θα μπορούσαν, εάν το ήθελαν, να βρουν πολλέ ε, δικαιολογίε για να τραβήξουν σε μήκο όλη αυτή την ιστορία. Δίνουμε λοιπόν το αποτέλεσμα, φέρνουμε το αποτέλεσμα και μέσα στις προθεσμίες. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να λέει κανείς ε, εγώ θα ήθελα κάτι παραπάνω, δεν είμαι ευχαριστημένος κτλ. Επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε να κάνουμε και με μια διαδικασία όπου έχει ήδη ξεκινήσει η διαβούλευση για τη νέα μεταρρυθμίση της ΚΑΠ. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Γι' αυτό καλώ και τον ε, Πρόεδρο και την ε, Γραμματεία να μεριμνήσετε παρακαλώ ώστε να ξεκινήσει το χέτερο δυνατό στα αρχές του επόμενου έτους το Όμνιμπους και η γεωργική μεταρρύθμιση. Ο κύριος Δες, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ και για τα επενδυτικά σας λόγια, για την ταχεία ολοκλήρωση των προσπάθειών αυτών πρέπει να επισημάνω βεβαίως και να μαυρώσω κάπως αυτή την εικόνα ότι είχαμε από την αρχή των ε, συνομιλιών ε, υποστεί την επίθεση και την κατηγορία ότι εμείς θα ήμασταν εκείνοι οι οποίοι σκοπεύαμε να καθυστερήσουμε, να φέρουμε σε ε, υπέρβαση των χρονικών ορίων την όλη διαδικασία και όμως αποδείξαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε γρήγορα, να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και πριν ακόμα από τους άλλους, πριν καν αρχίσει ο χειμώνας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και λυπάμαι που παρεμβαίνω, αλλά έχουμε κάποια διαδικαστικά στοιχεία που θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Γιατί πολλοί από εσά, αλλά και στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαίρονται για το αποτέλεσμα της συμφωνίας και την κρίνουν πολύ ενδιαφέρουσα και για τον γεωργικό κόσμο. Αλλά αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι έχουμε ακόμη πολλά στο διαδικαστικό επίπεδο. Έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε ακόμη εκεί. Και μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για κανονισμό omnibus ε, με πολλά στελέχη και πολλές, ε, πολλά σκέλη νομικά αφορούν τον προπολογισμό, το δημοσιονομικό κανονισμό μεταξύ άλλων. Εμείς στην Γεωργία εργαστήκαμε γοργά και άρτια με αυτόνομο τρόπο. Καταλήξαμε σε αυτή την πολιτική συμφωνία, αλλά για την εφαρμογή της συμφωνίας έχουμε κάποια διαδικαστική πρακτικά στάδια που θα πρέπει να περάσουμε και θα, δεν θα είναι εύκολο να γίνουν, να, ε, να υλοποιηθούν όλα αυτά τα διαδικαστικά βήματα. Καταρχήν, η αρχική μας πρόταση ήταν ότι αν όλα τα σκέλη της διαπραγμάτευσης ε, προχωρούσαν κανονικά, η αρχική μας ιδέα ήταν η, η συμφωνία που είχαμε στην Επιτροπή Γεωργία, ε, υποβάλλοντας σε ψηφοφορία. Είχαμε μάλιστα προγραμματίσει για μεθαύριο την ψηφοφορία για τις 9 του μηνός. Τελικά δεν θα γίνει αυτή η προγραμματισμένη ψηφοφορία, γιατί στην ψηφοφορία θα εγκρίναμε την ε, συμφωνία ώστε να την διαβιβάζαμε σε επιτροπές προϋπολογισμών και ελέγχου προϋπολογισμού για να τη συμπεριλάβουν στην γενικότερη συμφωνία και να τη διαβιβάσουν στην Ολομέλεια. Δυστυχώς είναι γνωστό και συμφωνούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία στα υπόλοιπα σκέλη, ιδιαίτερα για το δημοσιονομικό κανονισμό πριν τα τέλη του έτου. ή εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να γίνει τόσο γρήγορα ώστε να μπορέσει από την 1η Πρώτου του 2018 να τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός Omnibus. Εξού και η ιδέα που προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα και ταυτόχρονα ε, στους αρμόδιους για τη Γεωργία, στο Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσουμε σε αυτή τη διάσπαση, στο splitting που λέμε, στη διάσπαση, το διαχωρισμό αυτού των του κειμένου ώστε να διασφαλίσουμε, να διαφυλάξουμε αυτή τη γεωργική συμφωνία που στέκεται μια χαρά στα πόδια του προς το περιεχόμενο, να, να αφαιρέσουμε ε, αυτό το τμήμα από το, την αρχική πρόταση ώστε να προωθήσουμε την έγκριση και τη θέση ισχύ του με τη μορφή ενός ε, ξεχωριστού νομοθετικού μέσου του κανονισμού για την ε, ενδιάμεση εφαρμογή τη κοινή γεωργικής πολιτικής με άλλο τίτλο τέλο πάντων που θα αφορά όμω μόνο τη γεωργία. Και μάλιστα στι 12 Οκτωβρίου καταλήξαμε στη σχετική συμφωνία. Εκεί που περιπλέκονται τώρα τα πράγματα είναι ότι ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τα τέλη του έτου. Υπάρχει ένα πρόβλημα ακολουθίας, ε, λογικής ακολουθία ή αλληλουχία. Ποιο θα αποφασίσει για αυτή τη διάσπαση που έγινε τη πρόταση Omnibus. Η οι συνομοθέτε πρέπει να το κάνουν, δηλαδή το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την ΜΕΑ, από τη μόνιμη, Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διάσκεψη των Προέδρων είναι αρμόδια για τη λήψη τη σχετική απόφαση επί τη αρχή. Πώ θα γίνει κάτι τέτοιο έγιναν πολλές διαβουλεύσεις με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις υπηρεσίες των άλλων θεσμικών οργάνων και η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής. Ε, η διάσκεψη των Προέδρων ε, θα αποφασίσει υπό δύο όρους. Καταρχήν πρέπει να καλέσουμε την διάσκεψη των Προέδρων να λάβει την απόφαση και για να γίνει αυτό θα πρέπει να ε, συντάξουμε μία επιστολή που θα συνυπογράψουν και οι τρεις αρμόδιες επιτροπές, δηλαδή η κυρία Γκρέσλα και ο κύριο Αρτού από τι επιτροπέ προπολογισμών και Ελέγχου προπολογισμού και ο κύριο Εκέρς και ο Πρόεδρο τη Επιτροπή Γεωργία, Οι τρει πρόεδροι λοιπόν πρέπει να συνυπογράψουν την επιστολή που θα καλεί την διάσκεψη των πρόεδρων να λάβει τη σχετική απόφαση και η διάσκεψη των πρόεδρων δεν μπορεί να λάβει απόφαση, μα έχει ενημερώσει, παρά μετά την λήψη της απόφασης από το Συμβούλιο πρώτα. Οπότε πρώτα θα πρέπει η Κορεπέρ, η, μόνιμη, η Επιτροπή Μονίμων Επιτροσώπων να λάβει την απόφαση και μετά εμείς η διάσκεψη των Προέδρων. Ως προς το χρονοδιάγραμμα και αυτό έχει τροποποιηθεί γιατί υπάρχουν επιφυλάξεις από όλες τις πλευρές. Ε, με την τελευταία πρόταση για το χρονοδιάγραμμα φαίνεται ότι η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων 2 θα λάβει την απόφαση την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και ευελπιστούμε η Επιτροπή που δεν απαιτείται να αποφασίσει, αλλά καλό θα ήταν να στηρίξει αυτή τη διαδικασία, να επιβεβαιώσει και η Επιτροπή λοιπόν τη θετική της γνώμη με μια απόφαση που ελπίζουμε ότι θα εκδοθεί στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας. Οπότε, αν επιβεβαιωθεί αυτή η ακολουθία των γεγονότων, θα έχουμε λοιπόν την απόφαση της Κορεπέρ 2 στις 15 Νοεμβρίου και μετά έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Γιατί, Γιατί θέλουμε ε, να υιοθετηθεί το θέμα στη, το πακέτο, η συμφωνία του νέου αυτονομοθετικού οργάνου για την ε, γεωργική πολιτική στη Μήνη Ολομέλεια στις 29 και 30 Νοεμβρίου. Γιατί αν πάει στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, όχι απολύτως αδύνατο, αλλά πάρα πολύ δύσκολο και θα είναι τεράστιος ο κίνδυνος να μην προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι για την 1η Πρώτου 2018. Οπότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εγκριθεί αυτό το θέμα στη μήνυ ολομέλεια της 29ης και 30ης Νοεμβρίου. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει προηγηθεί στις 15 Νοεμβρίου η απόφαση της Κορεπέρ 2 κατόπιν. Ελπίζουμε στις 16 Νοεμβρίου την επόμενη Πέμπτη να αποφασίσει η διάσκεψη των ε, Προέδρων. Μάλιστα 10 το πρωί θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων. Κάνουμε ακροβατισμού εδώ. Ελπίζουμε στι 10 το πρωί η διάσκεψη των Προέδρων, 16 του μηνό, να αποφασίσει, ώστε ε, να υποβληθεί πριν το τέλο τη Συνόδου των, ε, την Πέμπτη να υποβληθεί αυτό το θέμα. Είναι δυνατόν παρά τον ακροβατικό χαρακτήρα του όλου εγχειρήματο και αν γίνουν όλα αυτά θα ε, υποβληθεί προς έγκριση το θέμα στην Ολομέλη 29 και 30 Νοεμβρίου ώστε να τεθεί να είναι έτοιμο για θέση εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Θα πρέπει όμως πρώτα το Κορεπέρ 2 να αποφασίσει στις 15 Νοεμβρίου όπως έχει αναγγείλει. Αυτά λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες. Και επίσης η δική μας η διάσκεψη των Προέδρων να λάβει την απόφασή της στις 16 Νοεμβρίου. Όλα είναι προγραμματισμένα με χειρουργική ακρίβεια. Επίσης, θα πρέπει προηγουμένως να στείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο Ταγιάννη, καλώντας την, Επιτροπή, την διάσκεψη των Πρόεδρων να λάβει να περιλάβει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και χρειαζόμαστε τις υπογραφές και της κυρίας Γκρέσλε και του κυρίου Αρτουή. Κάτι που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να συγκεντρώσουμε. Γιατί θέλουμε τις υπογραφές και των τριών αρμόδιων προέδρων. Είπα βέβαια ότι θα περιμένουν πρώτα την απόφαση της Κορεπερ 2, αλλά θα πρέπει να υπογράψουν οι πρόεδροι των Επιτροπών Προϋπολογισμών και Ελέγχου Προϋπολογισμού, Αρτουή και Κρέσλε και επίση να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη τη διάσκεψης των Προέδρων τη 16 η Νοεμβρίου. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, θα υλοποιήσουμε τον ποθετό στόχο να εγκριθεί δηλαδή το πακέτο στην Ολομέλη 29 και 30 Νοεμβρίου, στη Μήνη Ολομέλη, για να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018. Σα. λυπάμαι που σα κοράζω με όλε αυτές τι λεπτομέρειες, αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και κάνουμε πραγματικά φοβερέ ακροβασίε. Ε, προσπαθώντας να διασφαλίσουμε αυτή την τόσο καλή συμφωνία και τη θέση εφαρμογή της. Και νομίζω ότι αν δεν τεθεί αυτό από την 1η Πρώτου 2018 σε εφαρμογή, ε, θα αναβληθεί επαόριστον. Θα πάει για τις ελληνικές καλέδες, όπως λέμε, κάτι που δεν θα περιποιήσει τιμή σε κανένα θεσμικό όργανο. Εν πάση περιπτώσει κινητοποιηθείτε και ε, επικεντρώστε την προσοχή σας ε, στους προέδρους ε, Αρτουή, Γκρέσλε και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη, ώστε να προλάβουμε να τηρήσουμε όλες αυτές τις προθεσμίες και να φέρουμε σε αίσιο πέρα σε αυτό το πακέτο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Γραμματέφ, γιατί πραγματικά με τις εξηγήσεις μας διαφωτίσατε περί της διαδικασίας. Νομίζω όμως ότι είναι όλα θέμα πολιτικής βούλησης. Εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, όλα είναι δυνατά. Ε, το έχουμε διαπιστώσει και στο παρελθόν επανειλημμένος, ότι το κέριο ζήτημα είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης. Και φυσικά χρειάζεται και αυτή η επαφή με τους Προέδρους των άλλων δύο αρμόδιων επιτροπών, ώστε να καλέσουμε τη διάσκεψη των Προέδρων να λάβει τη σχετική απόφαση. Θα έχουμε λοιπόν την επαφή με την Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Είναι αρκετά περίπλοκη η διαδικασία, αλλά πιστεύω ότι είναι δυνατόν και εφικτό να επιτύχουμε το στόχο μας τηρώντας τη διαδικασία που μας περιέγραψε ο γραμματέας. Σας ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ τους κυρίους Ντές και Ντεκάστρο και ε, ευχαριστώ θερμά για την πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε και την επικοδομητική επίσης συνεργασία. Θερμές ευχαριστίες προς όλους και ευχαριστώ και την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλει κανείς άλλος το λόγο παρακαλώ από την Ομιγύρη. Ο κύριος γιάρμη πως; Όχι, κανείς άλλος. Οπότε επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου και πραγματικά να τις διαβιβάσετε και στον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή. Περνάμε στο επόμενο σημείο, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προώθηση των Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών και την ενθάρρυνση της παραγωγής πρωτεΐνης από ψυχανθή φυτά στον ευρωπαϊκό γεωργικό κλάδο. Αρμόδιος ε, εισηγητής είναι ο κύριος Δενανό. Θα θυμάστε την ακρόαση που είχαμε στην Επιτροπή μας με εκπροσώπους της ε, Ουγγαρίας και της Γερμανίας που μας παρουσίασαν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Σόγια. Η σχετική δημόσια ακρόαση είχε γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή μας και τότε ο εισηγητής, ο κύριος Πολ Ντενανό, μας παρουσίασε εκτενώς ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ελλείμματος που έχουμε στην ε, πρωτεϊνική μας παραγωγή. Ε, είχαμε εκτενή συζήτηση και στη δημόσια κρόση. Σήμερα θα έχουμε την ειδική εξέταση της έκθεσης Ντενανό, στον οποίο θα δώσω και το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Ο κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω αυτό το σχέδιο έκθεσης. στερα από πολλές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με εκπροσώπους της γεωργίας, των καλλιεργητών, των επιστημόνων. Προσπαθούμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα αυτό γιατί έχουμε σοβαρό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια στα πρωτεϊνούχες καλλιέργειες για τι ζωοτροφέ και το κοινοβούλιο έχει ασχοληθεί επανειλημμένω με το θέμα αυτό, επισημάνοντα ότι υπάρχει ανάγκη για, ένα σχεδιασμό, ε, ο οποίο όμω δεν έχει οδηγήσει σε πραγματική μείωση τη εξαρτησή μα από τι εισαγωγέ. Στο παρελθόν νομίζω η ανάλυση έχει γίνει μόνο από την οπτική των πρωτεϊνούχων ε, και το έλλειμμα το οποίο συμπληρώνουμε παγίως με εισαγωγές κυρίως σόγιας. Ωστόσο όμως τα πρωτεϊνούχα ως ε, γενικότερος προβληματισμός έχουν πολύ ευρύτερη πολύ ευρύτερες διαστάσεις ε, και έχουμε να κάνουμε και βέβαια με την ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου για την επάρκεια, την επάρκεια προμήθεια σε τρόφιμα αφενός, αλλά και την αντιμετώπιση του κινδύνου του κλιματικού ή περιβαλλοντικού. Έτσι λοιπόν οι εισαγωγέ ε, σόγιας έχουν, επηρεαστεί, έχουν επηρεαστεί σημαντικά από διακυμάνσεις τιμών ε, που εξαρτώνται βεβαίω από τη σημαντική αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο της ζήτηση, αλλά και τις δημογραφικές εξελίξεις και εδώ ιδιαίτερος κρούμε τον κόνο του κινδύνου σε σχέση με την Κίνα η οποία προτιμά τη δική της ε, επάρκεια προμηθειών σε σχέση με τους ε, λοιπούς, ε, συνάποντας ιδιαίτερες συμφωνίες με την Βραζιλία. Επίσης, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι επιτοπλίστων οι οργανισμοί, οι σπόροι σόγιας που εισάγονται, οπότε απορρίπτονται από την Ευρωπαϊκή αγορά εν γέννη. Επιπλέον, χρειάζεται για την καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων ε, εν γέννη φυτικών ε, ε, προϊόντων η κατανάλωση, η χρήση μάλλον μεγάλων ποσοστών αζότου με σημαντικές συνέπειες και για την ποιότητα των εδαφών αλλά και του, της ατμοσφαιρικής ποιότητας. Και γι' αυτό πρέπει να στραφούμε προς πρωτεϊνούχες καλλιέργειες που μπορούν να συγκρατούν τα ζωτούχα από το ατμοσφαιρικό αέρα και να βελτιώνουν ε, τον αέρα αυτό αντί να επιδεινώνουν την ποιότητά του. Χρειάζεται λοιπόν μια προσαρμογή στις ε, φυτικές πρωτεΐνες, αντικατάσταση των εισαγωμένων και μια προσαρμογή η οποία θα πρέπει να αποτρέψει τις ε, ανισορροπίες σε τοπικό επίπεδο ή την εξάρτηση σε παγκόσμια, από την παγκόσμια σκηνή. Μια βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν με μια σοβαρή ε, αναγνώριση της θέσης που έχουν οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τις σημασίες τους για τη μείωση της εξάρτησής μας από φυτικές πρωτεΐνες. Έτσι λοιπόν προτείνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα σχέδιο φιλόδοξο, ευρύ, για φυτικές πρωτεΐνες με αλλαγή, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, του σχεδίου παραγωγής, Ενό σχεδίου το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε διάφορους στόχου. πρέπει να ανταποκρίνεται, παραδείγματι, να εκδηλώνει ενδιαφέρον για όλους τους σπόρου και τις καλλιέργειες που είναι χρήσιμε για την ανθρώπινη ε, τροφική αλυσίδα αλλά και τις ζωοτροφές. Επίσης πρέπει να κοιτάξουμε τα όσπρια που μπορεί να έχουν ε, ενδιαφέρον είτε για τον άνθρωπο είτε για τις ζωοτροφές με πολύ μεγάλο αγρονομικό ενδιαφέρον. Παραγωγή επίσης βιομάζας στο μέγιστο θα πρέπει να μας απασχολήσει και για την ε, ανάπτυξη νέων πρωτεϊνών αλλά και για την εξασφάλιση κάλυψης των αναγκών κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης η παραγωγή θα πρέπει να έχει στόχευση εδαφική και να προσφέρει και νέες καλλιέργειες σόγιας με καλύτερα προσαρμοσμένες στις κλιματικές μας συνθήκες ε, ποικιλίε, άρα και καλύτερα αλλά και με άλλες ε, πρωτεϊνικές ή πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Και θέλουμε να στήσουμε βεβαίω την ε, προαγωγή των ψυχανθών και πρωτεϊνούχων, της μυδικής, του τριφυλιού, της τριτικάλη ζέας και πολλών άλλων αντίστοιχων καλλιεργειών. Έρευνε Βεβαίω θα πρέπει να γίνουν για την επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών, την προστασία, την ε, πεψιμότητα των καλλιεργιών αυτών από τον άνθρωπο αλλά και το ζώο, ε, προσαρμογή και ακρίβεια, ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από την φυτική αυτή παραγωγή και ώστε δυνατόν λιγότερη ε, σπατάλη, καλύτερη αντίληψη του κύκλου ζωής, ε, αμοιβεοποίηση των επιχειρήσεων ή ε, πειραμάτων και των γνώσεων που συλλέγονται και καλύτερη συνεργασία. Πρέπει μέσα κοινοτικά που μπορεί να έχουν συνέπεια στις καλλιέργειες των πρωτεϊνούχων να κινητοποιηθούν μέσα από τον πρώτο πυλώνα ήδη αυτό συμβαίνει σχέση με την ΚΑΠ με, την επιδοτήσει με τις ε, επιδοτήσεις, με τις ενισχύσεις για το πρασίνισμα, αλλά και για τις ε, πρόσθετες ενισχύσεις που θα πρέπει να, να διατηρηθούν αλλά και να ενισχυθούν. Επίσης έχουμε αγροπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το πρασίνισμα την, ε, μέσα στην διαδικασία της παραγωγής και επεξεργασίας αλλά και στη διαβίβαση της τεχνογνωσίας, την ενίσχυση των μικρομεσαίων την αξιοποίηση στην διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων, την αποτροπή των γενετικά τροπημένων οργανισμών. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε και ένα μείγμα καλλιεργειών και να εξασφαλίσουμε την προστασία και την ενίσχυση και για την ανάληψη κινδύνου όποιου ε, είναι διατεθειμένος να προωθήσει πρωτεϊνικές καλλιέργειες. Έρευνα, έρευνα που θα πρέπει να ενισχυθεί και από το κρατικό σκέλος απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Πολύ συχνά την έρευνα την αναλαμβάνουν ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι δεν έχουν σαν κύριο μέλημα παρά μόνο την αποδοτικότητα και όχι την ποιότητα. Επίσης, η πολιτική γειτονία έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να την ε, εξετάσουμε με προσοχή. Η Ουκρανία, Φερρυπίν, έχει ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες για την καλλιέργεια κυρίως της Όγιας. Η συνεργασία λοιπόν με την ε, Ουκρανία θα ήταν ίσως μια καλή λύση εν προκειμένου και θα μας επέτρεπε να ε, ασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε επαρκείς ποσότητες σόγες. Για την ε, ε, την πρωτεϊνούχα επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι οι συμφωνίες του Blair House του 1992 είναι πλέον ξεπερασμένες. Δεν αρκούν και δεν αντιστοιχούν και στις ανάγκες και τους κινδύνους από την κλιματική περιβαλλοντική αλλαγή. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αξιοποιήσουμε το όσο το δυνατόν ευνοϊκό πλαίσιο που έχουμε μετά την θετική δήλωση του Συμβουλίου και γενικά την, ε, τις ευνοϊκές συνθήκες για, τις, για τα πρωτεϊνούχα, να διατυπώσουμε την υποστήριξη μας στην έκθεση και την υποστήριξη προς τα πρωτεϊνούχα με μια επιφύλαξη βεβαίως ότι δεν μπορέσαμε να καλύψουμε σε αυτό το σχέδιο έκθεσης κάθε είδους ζήτημα ή ε, ερωτηματικό ή απορία σχετική με τα πρωτεϊνούχα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να, γίνει, να συνεχιστεί και η περαιτέρω συζήτηση και περιμένω να ακούσω τι έχει να πει η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντενανό. Θα ήθελα Τώρα να δώσουμε το λόγο στους και ηγητές ή στους αντικαταστάτες. Ο κύριος Λουαζό πρώτα. Oui, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή μας. Επιτέλους το να θεωρούμε ότι είναι ξεπερασμένη η συμφωνία του Blair House, όπως δήλωσε ο εισηγητή και ήταν ολέθρης από την αρχή, κάτι που καταγγέλουμε εδώ και πολλά χρόνια και μας κάνουν να υφιστάμεθα τις, τις συνέπειες ευρωπαϊκής, ε, στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Η Γαλλία ήταν από την αρχή κατά των, των συμφωνιών του Blair House. Χρειάστηκε όμως να υποκύψει και να τις εφαρμόσει τελικά επιτέλους γίνεται μια πρόταση για να θέσουμε ένα τέρμα στην εξάρτησή μας που οργανώθηκε με σε μεγάλο βαθμό και με την συνενοχή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ενθαρρυνθούν να παράγουν περισσότερους πρωτεϊνόχους, πρωτεϊνόχους καρπούς για να εξασφαλίσουμε μια πιστιστική αυτάρκεια. Αυτός είναι ο στόχος ήταν και ο στόχο, αλλά είδε το αποτέλεσμα σήμερα. Η εξάρτησή μα είναι μεγάλη. Θα καταθέσουμε τροπολογίε από την ομάδα μα στην ΕΝΕΦ και ελπίζω να γίνουν δεκτέ και να υπερψηφιστούν και από τις άλλες ομάδες. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία απ' όλα με ευχαριστήσω, Τόν. ή αλλως Ο κυριος χαιτεμα ναι, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Τόνισε νομίζω τα πιο σημαντικά σημεία αυτή τη έκθεση ήδη και πράγματι θα πρέπει να κοιτάξουμε στο μέλλον εάν μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας ε, από τις πρωτεΐνες τρίτων χωρών. Χαίρομαι λοιπόν που το συζητάμε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το συζητούσαμε εδώ και 15 χρόνια, αλλά απαιτείται κάποια δράση και πράγματι. Πρέπει να δούμε όχι μόνο τα πρωτεϊνούχα, αλλά όλους τους φόρους. Ε, γνωρίζω πως αυτή η έκθεση διασπρωτοβουλίας ε, δεν ασχολείται ειδικά με αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να πω στην Κομισιόν ότι μπορούμε να ζητήσουμε και άλλες πρωτεΐνες στα έντομα, αλλά και στις μεταποιημένες ζωτικές πρωτεΐνες που είναι ασφαλείς για ανθρώπινη κατανάλωση, κατηγορίας 3, πρωτεΐνες από το γρασίδι και, και το, τη χορτονομή και νομίζω ότι το σημαντικότερο εδώ πέρα είναι να αυξηθεί η απόδοση καλύτερη, καλύτερα υβρίδια και καλύτερες αποδόσεις και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε κάποια ασφάλεια για τους καλλιεργητές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην αναπαραγωγή και την καλλιέργεια νέων ειδών, αλλά χρειάζονται και μια βεβαιότητα ότι αν επενδύσουν θα έχουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο και μια βεβαιότητα ότι θα βγάλουν τα λεφτά τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα το πώς θα γίνει με την κοινή γεωρική πολιτική με άλλα μέση δεν το ξέρω, αλλά νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, όντως. το τελευταίο καιρό ίσως ε, παραμελήσαμε τις βελτιώσεις αυτών το, σε αυτό το είδος ε, των φυτών. Δίκιο έχετε. Ο κύριος Άγνιο. Thank you. Well, we're, we're talking about the item on the... agenda. Ευχαριστώ. Ε, συζητάμε το θέμα αυτό μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση των πρωτοεινούχων καλλιεργειών και υπάρχει μια δήλωση εδώ πέρα με την οποία δεν διαφωνώ. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη εξάρτηση από το εξωτερικό για τις πρωτεΐνες και μετά περνάει σε κάτι περιβαλλοντικά και λέει το εξής η χρήση των συνθετικών λιπασμάτων που περιέχουν άζωτο για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων έχει ένα φαινόμενο ντόμινο το οποίο μολύνει το νερό και παράγει ε, αέριο του θερμοκηπίου. Εδώ πέρα διαφωνώ γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι ψυχανθή. Φασόλια, λούπινα, τριφύλι κτλ. Όλα αυτά παράγουν το δικό τους άζωτο. Το παίρνουν από τον αέρα δηλαδή. Δεν χρειάζονται αζωτούχο. Ε. ούτε κλείουν κάποιο αέριο, αλλά εδώ πέρα δεν συνειδητοποιεί ο συντάκτης ότι προκαλούν ένα αέριο του θερμοκηπίου. Είναι βεβαίως ε, ένα αέριο το οποίο δεν έχει ουδέμια σχέση με το, οξύ, με το διοξίδιο του αζώτου. Πρέπει να σβήσουμε λοιπόν αυτές οι δύο αράδες εδώ. Δεν θα αλλάξουμε εδώ τον καιρό του κόσμου με τις καλλιέργειες. Η έκθεση αυτή τώρα μπαίνει πάρα πολύ στις λεπτομέρειες καλλιέργειας. Δεν χρειάζεται να μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πώς θα καλλιεργούμε πρωτεϊνούχα. Το, το μόνο που κάνουμε είναι να το δυσκολεύουμε με το να λέμε ότι δεν ε, πρέπει να έχουν ε, μέσα φυτοπροστασίας. Ε, δηλαδή βασικά βιολογική καλλιέργεια, δηλαδή τεράστια κίνδυνοι. Μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλο ποσοστό των ε, καλλιεργειών ψυχανθών είναι σπόρος και είναι πάρα πολύ ακριβά. Και αν βραχεί ή χαλάσει, έχει χάσει τα πάντα. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο βήμα Ουσιαστικά τους λέμε μην καλλιεργείτε πρωτεϊνούχα στις ε, περιοχές ε, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος γιατί ε, θα σας κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Και ο συνάδελφός μου εδώ πέρα λέει να αυξηθεί η απόδοση και να φέρουμε και τις σόγια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τι λέμε όχι, όχι, μην αγγίξετε τα γενετικά τροποποιημένα και επίσης και τα υβρίδια το ίδιο αυτά είναι γελία πράγματα. Αν ε, θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει κάποιους όρους για να υλοποιήσουμε, για να περιορίσουμε τα προβλήματα στον τρόπο τομέα αυτό. Κύριος Γιάρ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που καμιά φορά με ενοχλεί στην πολιτική δουλειά μας είναι ότι ο καθένα έχει το δικό του χώρο δραστηριοποίηση, ε, ζητάει αυτό που θέλει και δεν είναι τεθειμένος σε συμβασμού. Ε, σε αυτό θα ήθελα λοιπόν να συμπληρώσω ότι μπορεί πότε πότε να έχουμε κάποια σημεία τα οποία μας ενοχλούν, ειδικά στη στρατηγική για, την, ε, για τις πρωτεϊνούχες ε, καλλιέργειες. Η κράμβη πρώτα απ' όλα. Μπορεί βέβαια να μην ισχύει πάντα αυτό, αλλά από την κράμβη μπορούμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και βεβαίως κραμβέλαιο μπορούμε να εξάγουμε. Μιλούμε για ενέργεια πρώτης γενεάς. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι μαζί. Να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα. γιατί και το ε, κραμβέλο μπορούμε να έχουμε αλλά και ως παραπροϊόν της εξαγωγής του κραμβελαίου μπορούμε να έχουμε το πρωτεϊνούχο ως ζωοτροφή. Επίσης, έχουμε μιλήσει, έχει μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει δώσει μάλιστα και διάφορα ωφέλη προκειμένου να πρασινίσουν καλλιέργειες, να υπάρχει απαγόρευση, εξάλληψη των ε, φυτοπροστατευτικών ε, προκειμένου και να προστατευτεί το περιβάλλον αλλά δεν μπορούμε ταυτόχρονα να λέμε ότι δεν παράγουμε τη σόγια και δεν θέλουμε και να εισάγουμε σόγια και αυτό είναι πολύ κακό Στο χοιρινό, στην παραγωγή χειρίου κρέατος δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το ζώο, ο χείρος είναι παμφάγο και άρα μπορούμε να του δώσουμε πρωτεΐνου ζωοτροφή. Γιατί θέλουμε να το κάνουμε φυτοφάγο. Ας του δώσουμε και κρέα σε τελευταία ανάλυση. Δεν χρειάζεται να είναι φυτικής προελεύσεως η πρωτεΐνη που θα το ταΐζουμε. Αυτό πάλι λύνει ένα μέρος του προβλήματος. Στα βοηδή τώρα και τη γαλακτοπαραγωγή. Μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε εκτάσεις με πρωτεϊνού και σκαλλιέργειες που θα επιτρέπουν και την αξιοποίηση της πρωτεΐνης και την γαλακτοπαραγωγή. Βεβαίως, κατά πρώτο λόγο μας ενδιαφέρει το γάλα, αλλά ταυτόχρονα και το λιβάδι θα πρέπει να συντηρείται, να καλλιεργείται σωστά, να έχει και τα σχετικά φυτοπροστατευτικά ή τα λοιπάσματά του, και πάλι για κάποιους λόγους βλέπουμε ότι αυτά δεν επιτρέπονται από διάφορα περιβαλλοντικά ή άλλα προγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ας είμαστε λογικοί, δεν μπορούμε να έχουμε ακραίες θέσεις και τελικά να μην μπορούμε να φέρουμε κανένα αποτέλεσμα γιατί οι κερδισμένοι είναι από την άλλη μεριά του ωκεάτνου. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν λάβει το μήνυμα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και δει η ε, Βραζιλία, η οποία είδε ότι εμείς προχωρούμε στο greening, το πρασίρισμα και είπα, τι ωραία, ας αυξήσω την παραγωγή σόγιας. Είναι απλά λοιπόν τα στοιχεία, απλά και κλασικά. Δεν μπορούμε να τα λησμονούμε τα κλασικά, τις κλασικές ανάγκες, αλλά όπως είπα, κοιτάξουμε και παραπέρα. Και στα όσπρια και στην ε, κράμβη και στις ε, ε, δυνατότητες για αξιοποίηση των λοιπόν καλλιεργιών και των παραπροϊόντων τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Μποβέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι το πρώτο σχέδιο προτάσεως του εισηγητή βεβαίως είναι έχει σωστό προσανατολισμό και κατεύθυνση, αλλά θα επιμείνω στο εξή τρία. Πρώτον, η συμφωνία του Πλέρ House 1992 έρχονται σε μια χρονική στιγμή όπου γίνεται η διαπραγμάτευση και της ΚΑΠ αφενός και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου αφετέρου. Άρα είναι μια λογική συμβαστική λύση η συμφωνία του Blair House στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Αλλά είναι συμφωνία χωρίς ημερομηνία λήξεως. Απεριόριστης διάρκειας. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το πραγματικό πρόβλημα. Με ανώτατο όριο 5 εκατομμύρια ή κάτι περισσότερο των νεκταρίων που δικαιούται να ε, καλλιεργεί με πρωτεϊνούχα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε την ουσία αυτή και μέσα από την έκθεση βέβαια του κ. Τυρανό, αλλά ίσως και για τις άλλες συστήσεις που θα έχουμε στο μέρο σε επόμενες εβδομάδες, γιατί έχουμε τον προσεχή γύρω σε μερικές ε, εβδομάδες τον προσεχή γύρω λοιπόν του ΠΟΕ. Πρέπει να επανατεθεί το ζήτημα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτή την υποχρέωση. Δεύτερον, πρόβλημα εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί από το ίδιο στρατόπεδο ακούω και τους ωραίους ε, λόγους που ζητούν περισσότερη πρωτεϊνική παραγωγή και ισορροπία, αλλά υπάρχει και χώρα ταυτόχρονα, λεγόμενη κάτω χώρες, η οποία μαζί με τους Βραζιλιάνους ε, ε, κατασκευάζει τεράστια λιμάνια, τα χρηματοδοτεί. Και βέβαια αυτό πρόξενε το εξή πρόβλημα, ότι η Βραζιλία μετατρέπεται με μία μονοκαλλιέργεια ουσιαστικά, με τη λογική της μονοκαλλιέργειας που είναι καταστροφική και για το περιβάλλον της και για τους καλλιεργικές της και ταυτόχρονα βέβαια σημαίνει και τεράστια απερίμωση και αποψηλώς των δασών. Και επίσης, τρίτο πρόβλημα, η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και θα υπενθυμίσω για όσους δεν ήταν εδώ στην προηγούμενη βουλευτική περίοδο πως είχαμε αγωνιστεί για απλές μεθόδους την ε, φορά ως αγρονομικό μέσον που μας επιτρέπει και την επανεισαγωγή της, ε, των πρωτεϊνούχων, των πρωτεϊνικών καλλιεργειών και πιστεύω ότι η δουλειά που θα γίνει με όλα αυτά τα στοιχεία αλλά και με τις τροπολογίες που θα κατευθούν φαντάζομαι ε, θα οδηγήσει σε μια βελτίωση της πορείας και της προετοιμασίας για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριος Ντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Τζένανο για την έκθεση, για την πρότασή του. Πολλά είναι τα θετικά. Κάποια δύο σημεία βέβαια θα πρέπει να τα καλύψουμε τις τροπολογίες μας. Πάντως, εν γέννη, μπορώ να πω ότι η στρατηγική για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, έχει πάρει πλέον ε, κομικοτραγικές διαστάσεις και μορφή και περιορίζουμε τις αγωγές και καταστρέφουμε την εσωτερική καλλιέργεια. Γιατί 300.000 εκτάρια έχουν βγει με απόφαση του ε, επιτρόπου. Ε, ο ίδιος ο Υπουργός Γεωργίας της Τσεχίας ήρθε να μου πει ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. 300.000 εκτάρια που θα μπορούσαμε ε, με 100 μόνο ευρώ στο εκτάριο ως ενίσχυση να δώσουμε το κίνητρο για να προχωρήσουν αυτές οι καλλιέργειες με 30 δηλαδή εκατομμύρια ευρώ θα είχαμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η καλύτερη στρατηγική για, τις, για την κάλυψη των αναγκών μας σε πρωτεΐνες ε, ήταν ε, οι ενισχύσεις, η προαγωγή των πρωτεϊνικών καλλιεργειών. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υποστηρίζεται πλέον αυτό. Άλλωστε ξέρουμε ότι και για την φορά είναι, είναι χρήσιμες οι πρωτεϊνικές καλλιέργειες. Επίσης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος συζητεί την, ε, ε, τα ποσοστά ανάμιξης για τα καύσιμα και έχουμε στην Κραμβή 3,4 εκατομμύρια τόνους ε, ζωοτροφή απαλλαγμένη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που είναι περίπου το 1 τρίτο της παραγόμενης κράμβης. Άρα έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ε, ζωοτροφής που προκύπτει ως παραπροϊόν της κράμβης μαζί με το μέλι της κράμβης όπως λέγεται και αυτό αντί να το προωθούμε κάνουμε ακόμη εισαγωγές από την Άτια Αμερική. Ο γιος μου ίδιος, ο οποίος είναι καλλιεργητής, αποφασίζει να εγκαταλείψει ε, την καλλιέργεια της κράμβης γιατί μου λέει μπαμπά δεν μπορώ, δεν είμαι στη θέση να διαθέσω και να αξιοποιήσω επαρκώς τα προϊόντα αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να εγκαταλείπουμε αυτή την προοπτική για το μέλλον ε, επιβάλλοντας τόσο υψηλό κόστος ουσιαστικά και ε, τα λεπορία για τον καλλιεργητή. Επίσης από τις ε, καλλιέργειες, από τις εκμεταλλεύσεις που έχω εγώ ε, βλέπουμε ότι τεράστιο ποσοστό, 90% προχωρούν σε άμυψη σπορά. Γιατί λοιπόν να μην τις υποστηρίξουμε, γιατί να μην τις βοηθήσουμε να διατηρήσουν το έδαφος τους υγιές και γόνιμο. Πρέπει να κοιτάξουμε την εικόνα στο σύνολό τη. Ας μην κοιτούμε μόνο με μονομένες λύσεις ή προβληματισμούς. Πρέπει να δώσουμε γενικότερες λύσεις για την γεωργία. Βέβαια δεν βλέπω πολλές πιθανότητες να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον. Αλλά δυστυχώς στην Ευρώπη βλέπω να οπισθοδρομούμε την να προχωρούμε. Η κυρία Σλάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή περιέχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία και πράγματι πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την Ολλανδία. Έχω τρία συγκεκριμένα σημεία όμως ε, στο πρώτο θέμα για τα πρώτα πρωτεϊνούχα σόγια και λούπινα ε, δεν ξέρουμε αν υπάρχει πράγμα τόσο μεγάλη έκθεση αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το πριμ ε, ε, πρασινίσματος και το πώς θα διατηρηθεί εξίσου ελκυστικό αλλά βεβαίως και το τι θα γίνει με τη χρήση μέσων φυτοπροστασίας στις περιοχές οικολογικής προτεραιότητας αλλά αυτό ε, είπαμε ότι δεν το, είχαμε, δεν το κάναμε στην Αδία και πάλι βρίσκεται εδώ πέρα επιπλέον βλέπουμε για την, ε, το τι μπορεί να γίνει για τη διαφορά και την εξάρτησή μας ε, όσον αφορά τις καλλιέργειες αυτές από τον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως την σχέση που θα έχει με την ε, Συμφωνία για το Κλίμα και τις μεγάλες κλίμακας εισαγωγές από τρίτες χώρες και το πιθανό μπλοκάρισμά τους και το πώς θα μπορέσουμε έτσι να προωθήσουμε τις καλλιέργειες στην Ευρώπη. Αλλά Νομίζω ότι έχουμε εδώ πέρα μπλέξει πράγματα τα οποία δεν ε, κολλάνε μεταξύ τους γιατί χρειάζεται να έχουμε και κάποια διατροφική ασφάλεια για ανθρώπους ε, και για ζώα. Και τέλος ε, στην Ευρώπη επίσης έχουμε και κάποιες περιοχές οι οποίες ε, υποκαλλιεργούνται και θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν πολύ εντονότερα ή να παραμείνουν ε, βεβαίως ε, ακαλλιέργητες μέχρι να υπάρξει η απαραίτητη οικονομική ανάγκη αλλά πρέπει νομίζω να τις χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικότερα ευχαριστώ σας ευχαριστώ ο κύριος Φλάνναγκαν. Κάτι το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει την έκθεση είναι αυτό το 38%. Το 38% των ζωοτροφών που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πρωτοεινούχων και δεν θα έχουμε βεβαίως πάντα την εγγύηση αυτής της ε, παροχής και από την ε, περιβαλλοντική σκοπιά δεν έχει κάποιο νόημα να καλλιεργούμε κάποια πράγματα ε, να φέρνουμε κάποια πράγματα σε, με πλοία, να τα ταΐζουμε στα ζώα και μετά να εξάγουμε το τελικό προϊόν και να αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή. Κάτι πρέπει να κάνουμε, πολλά έχουν υποθεί, αλλά ένας ε, τομέας είναι το ότι δεν είναι όλες οι πρωτεΐνες ίδιες. Υπάρχει και θέμα ποιότητας, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη σόγια με πρωτεΐνη μπιζελιών. Δεν βλέπω πώς γίνεται αυτό, γιατί τα αμινοξέα των μπιζελιών δεν είναι τα ίδια με τις ε, σόγιας. Οπότε, αν μιλάμε για αντικαταστασή της σόγιας, θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι το οποίο θα έχει ανάλογα αμινοξέα. Και Είχαμε μια εξαιρετική παρουσίαση στην Επιτροπή μας, είχαμε ειδικού ε, επί των πρωτεϊνών που ήταν πολύ πιστικοί και κάποιοι από αυτούς ε, μίλησαν για την πώληση σόγιας, σπόρων σόγιας ε, τροποποιημένων και μη τροποποιημένων και μας είπαν ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε διαφορά στην στρεματική απόδοση και μα είπε γιατί δεν θα μπορούσαμε να καλλιεργούμε πολύ περισσότερο ισόγεια στην Ευρώπη και μάλιστα είπε ότι θα μπορούσε να είναι δυνατόν και στην Ιρλανδία. Απλά είναι θέμα παράδοση. Τέλο πάντων, το συζητάμε εδώ και 15 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένουμε άλλα 15 χρόνια γιατί όπως πάνε τα πράγματα τα επόμενα 15 χρόνια δεν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πρωτεΐνες. Πρέπει να κάνουμε κάτι και γρήγορα. Ο κύριος Ανδρέα. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Ντενανό για την εξαιρετική του δουλειά και την παρουσίαση. Γιατί διατυπώνει και τους στρατηγικούς και άρα και στρατηγικούς ε, γεωπολιτικούς ε, προβληματισμούς, δεν είναι βραχυπρόθεσμοι αλλά μέσω και μακροπρόθεσμη η μελέτη που μας παρουσιάσει, αν κοιτάξουμε παραδείγματι του τύπου των συμβάσεων που διαπραγματεύεται τώρα η Κίνα, είναι συμβάσει που θα διαμορφώσουν την κατάσταση της την επόμενη 15 ετία, 20 ετία και όπως λέει και ο κύριος Δυνανό. Έχει έρθει πια η ώρα, ύστερα από 10-20 χρόνια που το συζητούμε, να λάβουμε αποφάσεις και να στέσουμε θέσουμε σε εφαρμογή. Πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συγκεκριμένους όρους να εκφράσει αυτά τα ε, μελήματα και το περιβάλλον βεβαίως, όπως και άλλοι τομείς καλύπτονται. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό, αλλά ιδιαίτερα θα σταθώ στο κλίμα, ε, η οποία δεν είναι μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, είναι για τώρα, για σήμερα. Όταν λοιπόν λέγεται στην έκθεση ότι γίνεται έκθεση στην κινητοποίηση, γενική κινητοποίηση όλων των πηγών πρωτεϊνούχων και όχι μόνο των ε, καλλιεργιών των πρωτεϊνιών που προέρχονται από σπριαλά και των λοιπόν από χορτονομές ε, κτλ. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αμελήσουμε, έχει τεράστια σημασία και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε. Ευχαριστώ κύριος Εκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ το, να ευχαριστήσω τον κύριο Τυρανό, τον εισηγητή, για την πολύ σημαντική του έκθεση πρωτοβουλίας. Και θέλω, αγαπητοί συναδέλφοι, αγαπητές συναδέλφοι, να σας, ευχαριστώ, να σας υπενθυμίσω, Σκιώδης, εισηγητής ότι 10 20% της ε, σόγιας που καλλιεργείται από τον κόσμο πηγαίνει στην ανακατανάλωση από τον ανθρώπο, αλλά το 80% προορίζεται για ζωοτροφή πολύτιμη λοιπόν ε, παραγωγή και τροφή υποβαθμίζεται μετατρεπόμενη σε ζωοτροφή και ξέρετε ότι αυτό το έχω επισημάνει και κατακρίνει επανειλημμένος. Ε, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ε, για να έχουμε ζωική παραγωγή καλλιεργούμε την σόγια στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες και καταστρέφουμε τα τροπικά δάση παράγουμε αέρια θερμοκηπίου. Έμεσα βέβαια. Αυξάνουμε την παραγωγή ιδιαίτερα του μεθανίου λόγω των ε, εκπομπών από τα μυρικαστικά. Ε, ενισχύουμε τις ε, πιέσεις εις βάρος των ηθαγενών πληθυσμών της Νότιας κυρίως Αμερικής ε, και, τις εξα... και οδηγούμε στην εξάλληψή τους και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η χρήση της σόγιας ως ε, ζωοτροφής οδηγεί και σε τεράστια επιβάρυνση των υδάτινων αποθεμάτων του υδάτινου ορίζοντα. Λέγεται ότι στην Ευρώπη δεν είναι δυνατή αυτή η παραγωγή γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα της ε, διαφύλαξης των εδαφών και άρα εισάγουμε από την Ασία ή από τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Αλλά εμείς στην Ευρώπη, όσο και αν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε προσεκτικοί, έχουμε μεγάλη ευθύνη ακριβώς επειδή θέλουμε να τρώμε κρέας από τα ζώα. Έχουμε ευθύνη για την παραγωγή τη σόγια 35 εκατομμύρια τόνου το χρόνο και μα έχουν ξεπεράσει τώρα πια και οι Κινέζοι. Κάθε μέρα αυτό σημαίνει ότι εξαφανίζονται τεράστιες εκτάσεις στη Βραζιλία, την Αργεντινή και άλλες χώρες για την καλλιέργεια, υπέρ της της σόγιας και βέβαια αυτό επιβαρύνει και, το διοξίδιο, και σε διοξίδιο του άνθρακα την ε, ατμόσφαιρα της γης. Ε, είναι τεράστιες αυτές οι ποσότητες και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πρόκειται για σόγια γενετικά τροποποιημένη. Ο καταναλωτής στην Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει ότι χρησιμοποιούνται ζωοτροφές γενετικά τροποποιημένες. Είναι χρήσιμο λοιπόν το κείμενο αυτό, αυτή η έκθεση πρωτοβουλία και για να επενθυμίσουμε την ε, παραγωγή της σόγιας με γενετικά τροποποιημένο σπόρο και να ζητήσουμε αντί για αυτήν να προαχθεί η παραγωγή άλλων εναλλακτικών καλλιεργειών όπως της κράμβης και του κραμβελαίου στην Ευρώπη. Αλλά όπως είπα, μια καλή στρατηγική για τις ε, πρωτεϊνικές καλλιέργειες στην Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς αντίστοιχη στρατηγική και της μιας εισαγωγών στο σόγια αλλά και της κατανάλωσης κρέατος. Με αυτά θα βελτιωθεί και η δυνατότητά μας να επιτύχουμε τους μέσο και μακροπροθέσμους στόχους για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε πρωτοενικές καλλιέργειες δικές μας της Ευρώπης, εγχώριες, αλλά και ταυτόχρονα να αναλογιστούμε εάν θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Χρειαζόμαστε μια γεωργία πολύ πιο ε, ευνοϊκή ε, για το κλίμα, να μην οδηγεί σε κλιματική αλλαγή, που να μην είναι επιφερειμένη από γενετικά τροποποιημένη, που να μην είναι στραμμένη στα παγκοσμιοποιημένα, στα προϊόντα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Αυτά λοιπόν είναι τα δικά μου επιχειρήματα. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτά όλα να τα καταφέρουμε με την γενετικά τροποποιημένη σόγια που έρχεται από την άλλη όχθη του ωκεανού. Ο κύριος ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Ντενανό για τις προτάσεις που μας κάνει. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στον κανονισμό Omnibus ε, περιλάβαμε κάποια μέτρα ώστε να αντισταθμίσουμε τις απώλειες από το ε, ολέθριο μέτρο της, της απαγόρευσης χρήσης φυτοφάρμακων. Έτσι δίνουμε ε, κάποια όθηση και θα ρίνουμε τέτοιου είδους πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Οι πρωτεϊνικές καλλιέργειες στην Ευρώπη είναι κατεξοχήν καλλιέργειες ε, που εντάσσονται στην κυκλική οικονομία. Γι' αυτό και είναι εμβληματικό σχέδιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Γιατί με την παραγωγή κτηνοτροφικών πιτών αλλά και με τα έλαια που παράγονται για τους πλακούντες ε, για τα κτηνοτροφικά δηλαδή αυτά ε, τρόφιμα, χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τέτοια πρωτεϊνούχα. Επίσης, να μην ξεχνούμε το θέμα της έρευνας ε, γιατί και για τα αγροστόδη και για τα κτηνοτροφικά φυτά ε, οι έρευνες ε, τα τελευταία 30 χρόνια συνέβαλαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας αλλά λόγω της αδυναμίας των αγορών ο τομέα των πρωτεϊνούχων δεν βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας. Δεν υπήρχαν αρκετές επενδύσεις στην έρευνα για τα πρωτεϊνούχα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δίνουμε τις προσπάθειές μας γιατί χρειάζονται κρατικά κονδύλια ώστε τα ελαιούχα και τα πρωτεϊνούχα, κυρίως τα πρωτεϊνούχα στην Ευρώπη, να ε, λάβουν την δέουσα υποστήριξη, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι στιγμής. Ό,τι αφορά τα, τη σόγια, όντω. Ε, πριν από 30 χρόνια δεν είχαμε καθόλου σόγια. Χάρη στι ερευνητικέ προσπάθειε που έγιναν στις ποικιλίε έχουμε σήμερα ευρωπαϊκή σόγια, αλλά για τι άλλε ποικιλίε που αναφέρθηκαν ή μάλλον τα άλλα είδη, για παράδειγμα μυδική, λούπινα κτλ. Εκεί θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε αυτά τα φυτά και να τα προσαρμόσουμε στα εδάφη και τα κλίματα των χωρών μας γιατί πιστεύω ότι τέτοιου είδους ψυχανθή θα χρησιμεύσουν ιδιαίτερα στην αμύψη σπορά στην Ευρώπη και θα αποτελέσουν ένα πολύ ωφέλιμο σκέλος αυτής της αμύψης σποράς. Σας ευχαριστώ. Ε, εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομίλητων. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, παρέβλεψα την κυρία Μαγκίνες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την επίοικιά σας και ζητώ συγγνώμη από τον εισηγητή και τους συναδέλφους γιατί έφτασα καθυστερημένα. Λυπούμε. Ε, σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Νταντέ για την έρευνα. Το πρόβλημα με την πρωτενική προμήθεια στην Ευρώπη είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε πια ε, ε, κρεατάλευρα και οστεάλευρα στην Ευρώπη, χάνοντας έτσι μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης. Θα πρέπει στο εσωτερικό μας να αυξήσουμε την ε, προμήθεια πρωτοτεϊνούχων γιατί η Κίνα έχει αυξήσει την ε, κατανάλωση, την εισαγωγή σόγιας και δεν την ενδιαφέρει αν είναι γενετικώς τροποποιημένη ή όχι. Ή λοιπόν θα χρειαστεί να ε, ενδώσουμε στην γενετικώς τροποποιημένη σόγια ή να αυξήσουμε την ντόπια πρωτεϊνική παραγωγή. Επίσης, το σύστημα της προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης λειτουργεί μεν, αλλά πολύ περιορισμένα. Χρειαζόμαστε περαιτέρω κονδύλια στο τομέα αυτό για να στηρίξουμε την παραγωγή πρωτεϊνούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μια τέτοια στήριξη θα φέρει και πάλι το θέμα στο επίκεντρο τη προσοχή, Η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε μια σχετική στρατηγική και συμφωνώ με τον κύριο Ταντά ότι θέλουμε ε, επενδύσεις, ε, δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, γιατί οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν χρηματοδοτούν τέτοιου είδους έρευνα. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τενανό για την έκθεσή του και να υποσχεθώ ότι θα καταθέσω ένα μικρό αριθμό τροπολογιών. Ελπίζω να τις δεχτεί. Ε, κύριε Πέτυρε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό όντω είναι εξαιρετικά σημαντικό και είχαμε οργανώσει και στην Επιτροπή μας σχετική δημόσια ακρόαση όπου πυρογνώμονες από διάφορα ευρωπαϊκά Ινστιτούτα επιβεβαίωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει αυτάρκεια στην πρωτεϊνική της παραγωγή και στην, στις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές. Και ε, επίσης θέλουμε να μειώσουμε την εισαγωγή γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ιδιαίτερα τις σόγιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που όπως είπαμε η Κίνα δεν ενδιαφέρεται γιατί την ενδιαφέρει μόνο η εισαγωγή σόγιας. Επίσης ε, έχουμε μια ειδική ποικιλία σόγιας, τις σόγιας του Δούναβη ε, και μάλιστα και η Κροατία άρχισε να καλλιεργεί μη γενετικώς τροποποιημένη σόγια. Οπότε μπορούμε να εξασφαλίσουμε παραγωγή σόγιας που θα ε, καλύπτεται από έγκυρα πιστοποιητικά για μη γενετική τροποποίηση και πιστεύω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τέτοια παραγωγή ώστε να φτάνουν στο τραπέζι των καταναλωτών μας προϊόντα και τρόφιμα που θα έχουν πιστοποιητικό τροφίμων απαλλαγμένων από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Έχουμε τη δυνατότητα στην περιοχή γύρω από το Δούναβι να παράγουμε ε, μη γενετικώς τροποποιημένη σόγια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζονται όμω χρηματοδότηση και υποστήριξη τέτοιου είδου παραγωγή μη γενετικώς τροποποιημένη, γιατί είναι δεδομένο ότι είναι απολύτω απαραίτητη για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τώρα πραγματικά έχουμε ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών. Και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Γιένς Σχάπς, τον οποίο καλωσορίζουμε μαζί με τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Σχάπς έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Ντενανό για αυτή την έκθεση και την πρωτοβουλία. Για μας είναι σαφές ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει την δυνατότητα να βελτιώσει την χώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ε, πρέπει να στηριχθεί από την Κομισιόν. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουμε στο τωρινό πλαίσιο ε, της ε, κοινής πολιτικής κάποιες επιτυχίες από το 2013 έχουμε την εθελοντική στήριξη, η οποία άλλαξε κάπως το καθεστώς σε σχέση με το παρελθόν και ειδικά για την σόγια αλλά και για τα φασόλια, λούπινα και μπιζέλια είχαμε μια αύξηση των τελευταίων 5 ετών της εγχώριας παραγωγής κατά 15%. Οπότε το 2017 αναμένουμε ένα επίπεδο παραγωγής γύρω στο 2,7 εκατομμύρια τόνους σόγιας και 5,3 εκατομμύρια τόνους ε, ψυχανθών, κάτι το οποίο είναι συγκρίσιμο με το... κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το παρελθόν. Του τελευταίντος είναι σαφές ότι ε, με αυτό το επίπεδο δεν καλύπτουμε τις ανάγκες ε, που έχουμε στην Ευρώπη και ειδικά το έλλειμμα των πρωτεϊνούχων είναι πολύ υψηλό για τα πρωτεϊνούχα τα πολύ πλούσια όπως ε, η σόγια. Η σόγια είναι πολύ σημαντική γιατί ε, είναι ένα πολύ καλό προϊόν ε, για τις ζωοτροφές και γνωρίζουμε ότι η σόγια από σκοπιές πρωτεϊνών είναι πολύ σημαντική. Οπότε θα ήθελα να θα θέλαμε να δοθεί βάρος στην έρευνα στην γεωργία ακριβίας και βεβαίως μπορούμε να προσαρμοστούμε πολύ καλύτερα και στις κλιματικές συνθήκες της Ευρώπης. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι στο πλαίσιο του κανονισμού Omnibus είχαμε μια ξεκάθαρη δήλωση από τις υπηρεσίες της Κομισιόν επαναβεβαίωσουμε την πρόθεσή μας να ξαναδούμε την κατάσταση της προσφοράς και της ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να θαρρύνουμε περαιτέρω την παραγωγή πρωτεϊνούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο που θα στέκει οικονομικά και περιβαλλοντικά. Νομίζω αυτά επιβεβαιώνουν την δέσμευση της Κομισιόν για να υποστηριχθεί η παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών. Οπότε αναμένουμε την περαιτέρω συνεργασία με τον κύριο Ντένανο και την Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, το λόγο έχει ο συγκεκριτής μας ο κύριος Ντενανό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Νομίζω ήταν πολύ κατατοπιστική αυτή η συζήτηση και πραγματικά εντοπίστηκαν πολύ σημαντικά σημεία που θα εμπλουτίσουν την έκθεσή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χέιτεμα για την ιδέα του να δώσουμε εχέγγυα στους ε, Γιώργους, οικονομικά, γιατί ε, αν τους εθαρρύνουμε να παράγουν ψυχανθή θα πρέπει να δώσουμε κάποιες οικονομικές εγγύησεις. Ε, επίσης, ε, κύριε Άκνου, δεν κατάλαβα και πολύ καλά από αυτά που είπατε, γιατί είπατε ότι ε, τα ψυχανθή είναι αζωτοδεσμευτικά φυτά και άρα δεν χρειάζονται πολλά ζωτούχα λοιπάσματα. Συμφωνώ. Επίσης, οι ελαιοκράμβοι πολύ συχνά είναι ε, συμπροϊόν, όχι δηλαδή μόνο για την παραγωγή κτηνοτροφικών πρωτεϊνών, αλλά και για την παραγωγή βιομάζας. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Πετήρ ε, και με τους ε, άλλους συναδέλφους συμφωνώ και περιμένω τις τροπολογίες τους. Κύριε Ντές, μας υπενθυμίσατε τις συνολικές και τις μικτές καλλιέργειες, τις, το συνδυασμό καλλιέργειων. Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα, στην πολυμορφία των εδαφών μας, αλλά και στην ποιότητα και την πολυμορφία του κλίματός μας. Έτσι μπορούμε να παράγουμε πολύ περισσότερα πρωτεϊνούχα φυτά και να εξασφαλίσουμε μια αυτάρκεια. Σε ό,τι αφορά τους γενετικώς τραποποιημένους οργανισμούς, κυρίως τα πρωτεϊνούχα δεν πρόκειται με γενετικώ τροποποιημένους οργανισμού να λύσουμε το πρόβλημα της εξάρτησή μας ε, για πρωτεϊνούχα φυτά. Θα πρέπει να εξετάσουμε και αυτό το θέμα και είναι ευπρόσδεκτες σχετικές τροπολογίες. Κύριε Φλάναγκαν, επιβεβαιώνω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των αμινοξέων των ε, διαφόρων ε, φυτικών πρωτεϊνών. Σίγουρα η πρωτεϊνική απόδοση της σόγιας ε, είναι πολύ υψηλή, αλλά και άλλα φυτά όπως οι ελαιοκράμβοι έχουν υψηλό πρωτεϊνικό δυναμικό. Επίσης και κάποια γροστόδη ή κάποια πόδι ή χορ... καλλιέργειες χορτονομής προσφέρουν υψηλό επίπεδο πρωτεΐνης και ακόμη και είναι μικρές οι ποσότητες, ε, δεν θα πρέπει να τις αμελούμε ανάλογα με το κλίμα, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του εδάφους. Πιστεύω ότι κάθε χώρα, κάθε έδαφος, κάθε κλίμα μπορεί να συμβάλλει ε, στο να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε την εξάρτησή μας από την εισαγωγή πρωτεΐνης. Κύριε Εκ, όπως λέω και στην έκθεσή μου, θα πρέπει να αποκλείσουμε τις, τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, έστω και φτάνουν μέσω ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ζωοτροφών. Βέβαια είναι ένα μακρόπνο έργο, θα πρέπει να συνεχίσουμε πάντως τις προσπάθειες. Κύριε Νταντά, σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Όντως, το θέμα της κυκλικής οικονομίας είναι πολύ σημαντικό και δεν θα πρέπει να το αμέλουμε, θα πρέπει να το υπεθυμίζουμε συνεχώς. Επίσης, επισημαίνω στην έκθεση ότι είναι πολύ σημαντικό σημαντικό το θέμα των δημοσίων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της έρευνας, γιατί χωρίς τέτοια κρατικά κονδύλια για την έρευνα θα έχουμε πολύ ιδιωτικές έρευνες, πολύ τοπικά περιορισμένες που δεν θα ωφελούσαν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συμφωνώ κυρία Μαγκίνης για το θέμα της ε, έρευνας. Κυρία Πετήρ, μιλήσατε για το, το Δούναβι, την περιοχή γύρω από το Δούναβι και τις χώρες γύρω από το Δούναβι. Ε, και την σόγια. Όντως μπορεί αυτή η περιοχή και η παραγωγή στις χώρες αυτές μπορούν να συμβάλλουν στον αγώνα μας για τον περιορισμό της εξάρτησής μας από τις εισαγόμενες πρωτεΐνες. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμώ ιδιαίτερος ότι ε, ε, είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά και προσέχει τις προτάσεις και της δικής μας Επιτροπής και σίγουρα δεν θα πρέπει να μένουμε σε αβεβαιότητα γιατί η Βραζιλία θα υποστεί πολλά δεινά από τις συμφωνίες αυτές με την Κίνα. Και αν ε, η Βραζιλία κατακλείσει ε, την αγορά της Κίνας, οπότε δεν θα μπορέσει πια να εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα αντιμετωπίσουμε και εμείς πολύ σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι αυτό από καινού, μαζί με το Συμβούλιο, ώστε το θέμα των πρωτεϊνούχων να αποτελέσει μεγάλη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για τη γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για το σύνολό της και για τους πολίτες της. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι πραγματικά συζητήσαμε πολύ διεξοδικά αυτό το θέμα. Είχαμε όλοι το χρόνο να μιλήσουμε. Μέχρι 14 Νοεμβρίου στη μία το μεσημέρι παρακαλώ να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας γίνει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα με την σύμφωνη γνώμη της συντάκτριας της γνωμοδότησης της κυρίας Βιωρίτσα Νταντσίλα, δηλαδή το σημείο 7 ε, να βάλετε για λίγο αργότερα και θα περάσουμε πρώτα στο σημείο 8, την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Διευθύντη τον κύριο Κλάρκ, ε, του θέματος για την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα γιατί όπως ξέρετε κυρίως θέμα των συζητήσεων στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου είναι η προετοιμασία της 11ης Υπουργικής Διάσκεψης στον ΠΟΕ που θα λάβει χώρα 9 με 13 Δεκεμβρίου ε, με συμμετοχή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα συμμετέχουν ε, μεταξύ άλλων και η κυρία Μαγκίνες από την Επιτροπή Γεωργίας. Και μάλιστα η κυρία Μαγκίνες που είναι ταυτόχρονα και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα βοηθήσει πολύ στο να δοθεί το απαραίτητο βάρος ε, στην ε, παρουσίαση της θέσης μας, της Επιτροπής Γεωργίας. Για τα γεωρικά ζητήματα στον ΠΟΕ θα μας μιλήσει ο κύριος Κλάρκ. Και τον παρακαλώ να μην αμελήσει να μας παρουσιάσει και τις συνέπειες από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλήσει για τις δασμολογικές ε, ποσοστώσεις για το καθεστώς φυσικά του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΠΟΕ μετά το Brexit και τις πιθανές συνέπειες για τις υπόλοιπες 27 χώρες και για τις άτυπες συζητήσεις που ήδη έγιναν στη Γενέβη. Παρακαλώ κύριε Κλάρκ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως μου ζητήσατε θα κάνω την παρουσίαση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τη γεωργία στον ΠΟΕ εν ώψη της MC11 της ε, Υπουργικής Διασκέψης στην Αργεντινή και πολύ ευχαριστώ να απαντήσω και στις ερωτήσεις που ενδεχομένω να αφορούν και άλλα θέματα. Για να μην ε, σας ε, κουράσω με την πολυτεχνική παρουσίαση και να σταθώ κυρίως στα πολιτικά ζητήματα, θα ήθελα να αφορθώ και στα όσα συμβαίνουν στην ίδια αλλά και τι συνέπειες μπορεί να έχουν στην ισχύουσα ΚΑΠ, αλλά και το μέλλον της. Και θα σταθώ στο ερώτημα εάν ο ΠΟΕ μπορεί να περιορίσει την, ε, τη βάθμο ευελιξία που έχουμε είτε τώρα είτε στο μέλλον στην ΚΑΠ. Πώς βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΠΟΕ. Με δύο λόγια, μας θεωρούν αξιόπιστους, επικοδομητικούς, Υποστηρίζουμε την πολυμερή διάσταση των συνομιλιών και συμφωνιών. Είναι ήδη πολυμερής οργάνωση η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδια. Για δε τη γεωργία, ύστερα από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ, δεν βαλόμεθα πλέον και μάλιστα μπορέσαμε και να ηγηθούμε πριν από δύο χρόνια στο Ναϊρόμπι της πλήρους εξάλληψης των εξαγωγικών επιδοτήσεων, πράγμα αδιανόητο πριν από 5 ή 10 χρόνια ακόμα. Οι αλληλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ βεβαίως λαμβάνονται για λόγους εσωτερικής πολιτικής. Δεν έχουμε καλή πολιτική λόγω των οικονομικών συνθήκων. Αλλά με τις αλλαγές αυτές που επιφέρουμε στην ΚΑΠ ταυτόχρονα δεν πρέπει και να λησμονούμε τις, ε, τον αντίκτυπο του ΠΟΕ ή στον ΠΟΕ σε νομικό ή πολιτικό επίπεδο και εδώ ακριβώς δεν θέλω να σταθώ στην παρουσίασή μου. Η ενδεκάτη λοιπόν η Υπουργική Διάσκεψη θα γίνει στον Buenos Aires τον Δεκέμβριο. Κάθε δύο χρόνια είναι οι υπουργικές διασκέψεις του ΠΟΕ. Εδώ θα συζητηθούν και θα γίνει διαπραγματεύση για νέους πράσινους κανόνες και για, τον περαιτέρω, για την περαιτέρω πορεία. Τι προβλέπετε λοιπόν ως θέματα, πολλά έχουν συζητηθεί. Ε, στη Γεωργία θα είμαστε κυρίως εστιασμένοι στις επιδοτήσεις για την αλληλεία δηλαδή κανόνες για τον περιορισμό του όγκου των επιδοτήσεων που οδηγεί σε υπεραλίευση και βέβαια και ένα πακέτο για τα θέματα της γεωργίας. Τέσσερα κυρίως Θα απασχολήσουν τους υπουργού σε θέματα γεωργίας. Δημόσια συμμετοχή, αποθεματοποίησης, η υποστήριξη με τις ενισχύσεις ουσιαστικά της παραγωγής, κανόνες για το βαμβακά που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ε, βαμβακοπαραγωγούς χώρες της Δυτικής Αφρικής και περιορισμούς ή απαγορεύσεις ε, εξαγωγών. Αυτά είναι τα θέματα για τον Πόνος Άιρες. Ιστορικές ενισχύσεις καταρχάς, που είναι το πιο σημαντικό. Σε αυτό θα σταθώ κυρίως. Και ίσως και το θέμα το πιο άμεσα σχετιζόμενο με την ΚΑΠ και τον εξυγχρονισμό της στο μέλλον. Και προς τώρα τα κυριότερα μέλη της ΚΑΠ, τώρα είναι μελλοντικά, έχουν ένα ανώτατο επίπεδο δαπανών σε επιδοτήσεις στρεβλώσεως ανταγωνισμού. Είναι το λεγόμενο Amber Box, κίτρινο κουτί. Ε, όπως και οι άλλοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα περιθώριο από το Amber Box με τις δαπάνες που επιτρέπονται σε επιδοτήσεις. Ε, όπως και τα μέλη μας, οι κράτη-μέλη δηλαδή, δεν επιτρέπουμε να ξεπεράσουμε, να εξαντληθεί μάλλον αυτό το ποσό, αλλά και άλλα κράτη, Βραζιλία, Περού, Κολομβία, μαζί με μας έχουν προτείνει τον περιορισμό του όγκου της δαπάνης στην οποία μπορούν να προβούν τα κράτη με αυτό το amber box, δηλαδή τις λεγόμενες τρευλωτικές, τρευλωτικού αποτελέσματος ενισχύσεις. Θέλουμε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο αυτό το ποσό. Και αυτό το το επίπεδο, το βάνη θέλουμε την οροφή αυτή, θέλουμε να την ορίσουμε κατά τρόπον ώστε να μην περιορίσουμε τα τωρινά μας επίπεδα δαπανών, που είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία δικαιούμεθα με το τωρινό Amberbox. Εδώ λοιπόν έχουμε την πιο στρεβρωτική των εμπορικών συναλλαγών μορφή ενίσχυση στη γεωργία. Ταυτόχρονα όμω και αυτή είναι και η πρότασή μα στον ΠΟΕ, θα είμαστε διατεθειμένοι σε μια δεύτερη φάση να ε, ανοίξουμε και το λεγόμενο blue box, το μπλε κουτί, εφόσον πάντα ε, μένει περιθώριο και στην τωρινή και στην μυρωδική ΚΑΠ για διατήρηξη των δαπανών του Blue Box, το οποίο υποστηρίζει παραδείγματι το Βάμβακα στην Ελλάδα και την Ισπανία, ε, την κτηνοτροφία αλλά και κάποιες συγκεκριμένες καλλιέργειες σε μεταβαλλόμενα επίπεδα κτλ. Και τρίτον, προτείνουμε, μάλλον επιμένουμε στο ότι η αδίποτε μεταρρύθμιση και οι δίποτε κανόνες δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στο green box, το πράσινο κουτί που έχει να κάνει με τις άμεσες ενισχύσεις και τα προγράμματα ενίσχυσης του, της υπαίθρου. Αυτά λοιπόν θεωρούμε και επιμένουμε ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν πως τρευλώνουν τον ανταγωνισμό γιατί δεν ενισχύουν την παραγωγή. Άρα έχουμε φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, συνεχίζουμε στις στην προοδευτική αναθεώρηση της ΚΑΠ μας, ταυτόχρονα όμως αφήνουμε και περιθώριο για την ενίσχυση, για τη διατήρηση των ενισχύσεων και τώρα και στην προσεχή εκδοχή της ΚΑΠ. Άλλοι θέλουν να καταργηθούν τελείω οι ενισχύσει για όλου του παραγωγού. Δεν το θεωρούν ρεαλιστικό. Ούτε εμεί, ούτε και οι περισσότεροι από τα μέλη του ΠΟΕ. Και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βραζιλία αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να ενώσουν τι δυνάμει του σε μια κοινή πρόταση, νομίζω αντικατοπτρίζει και το γεγονό ότι έχουμε αλλάξει, έχει αλλάξει η ΚΑΠ. Είναι πιο σύγχρονη ε, και ανοιχτή σε λύσεις κοινέ με χώρες όπως η Βραζιλία. Και τώρα θα ήθελα να, σα να σας εξηγήσω τι σημαίνει συγκεκριμένα στην πράξη η πρότασή μας. Αν το βλέπετε... Πρόκειται για έναν πίνακα στον οποίο οι μπλε στήλες δείχνουν ε, το πόσο μας ε, επιτρέπεται να ξοδέψουμε σε στηρίξεις οι οποίες τρευλώνουν το εμπόριο ως ποσοστό της αξίας παραγωγής. Έχουμε μια αξία παραγωγής σε λίγο πάντα από τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας επιτρέπεται ένα 30% αυτής της αξίας, γύρω στο 110 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν. Στην πράξη ξοδεύουν ένα κλάσμα αυτού κάτω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ οπότε έχουμε αρκετά μεγάλο περιθώριο και προτείνουμε να μειωθεί ε, αυτό το πλαφόν αρκετά. Ναι, αν παραδείγματος χάρη βάζαμε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο, ας πούμε στο 15% της ε, αξίας της ε, παραγωγής θα κόβαμε έτσι όλο το περιθώριο αλλά δεν ε, θα υπήρχε πρόβλημα στην ε, καθημερινή ε, στην καθημερινή μας λειτουργία και δαπάνες. Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους πάντες με τρόπο σχετικά δίκαιο και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε δίκαιη μεταχείριση όλων των μελών του ΠΟΕ. Δηλαδή ότι ισχύει για μας, να ισχύει για Καναδά, Ιαπωνία, ΙΠΑ, Κίνα και λοιπούς. Αυτό δεν θα μείνω σε αυτό. Είναι μια ανάλυση του πώς ε, μετακινηθήκαμε από ενισχύσεις ε, που στρεβλώνουν ε, το εμπόριο, το καφέ και το μπλε. Ε, βλέπετε ότι σύν το χρόνο το έχουμε μειώσει και τώρα είμαστε όλοι στο πράσινο κομμάτι ανάπτυξη της υπαίθρου και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν κάνει ουσιαστικέ μεταρρυθμίσεις. Και βλέπετε κάπως διαφορετικά το πώς ξοδεύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων στην κοινή γεωργική πολιτική. Και βλέπουμε εδώ πέρα το πορτοκαλί κουτί είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια, το μπλε κουτί 5 δισεκατομμύρια και όλα τα υπόλοιπα είναι σχεδόν το πράσινο κουτί 38 δισεκατομμύρια το έτος ε, ε, κατά το οποίο περιλαμβάνει και την συγχρηματοδότηση των κρατών μελών. Οπότε, για να συνοψίσω, προτείνουμε μία περαιτέρω σταδιακή ε, μεταρρύθμιση των ενισχύσεων ε, θα συνεισφέρουμε και εμείς και άλλα μέλη που βρισκόνται σε παρόμοια κατάσταση αλλά θα έχουμε και αρκετό περιθώριο για να μειώσουμε το μπλε και το πράσινο κουτί στο μέλλον όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να στραφώ στο δεύτερο σημαντικό ζήτημα για την γεωργική ατζέντα μας και αφορά την δημόσια συμμετοχή. Αυτό αφορά κάποια συστήματα της Ινδίας και άλλων που αγοράζουν κάποια βασικά τρόφιμα, ρύζι, στάρι κτλ. Επιδοτώντας και την τιμή, πολύ ψηλότερα από την τιμή αγοράς και μετά αποθηκεύουν τα δημητριακά αυτά και τα μοιράζουν στους φτωχούς. Αφενός ε, είναι ένα θέμα θεμητό διατροφικής ασφάλειας, από την άλλη επιδοτούνται οι αγρότες με στήριξη των τιμών. Και αν μετά γίνει εξαγωγή αυτών των αποθεμάτων έχουμε στρέβλωση για τις άλλες χώρες πως ε, χώρες όπως οι Φιλιππίνες, το Πακιστάν και τα λοιπά ανησυχούν πολύ γι' αυτά πριν από τέσσερα χρόνια στο Μπαλί συμφωνήσαμε μια ενδιάμεση λύση για την Ινδία ε, στην οποία θα επιτρεπόταν να διατηρήσει αυτά τα συστήματα χωρίς ε, να μετράνε στο πορτοκαλί κουτί αλλά είπαμε ότι θα πρέπει να βρεθεί και μια μόνιμη λύση μέχρι το Buenos Aires τον επόμενο μήνα. Τα τρέχοντα λοιπόν συστήματα τα οποία εγκρίθηκαν προσωρινά από τον ΠΟ καλύπτουν τα παραδοσιακά αυτά προϊόντα, ρύζι και στάρι. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν από εδώ και μπρο. Θα επιτρέψουμε να συνεχιστούν όσο ε, έχουν αυτά τα συστήματα ή θα επιτρέψουμε ναι, την εισαγωγή νέων συστημάτων από νέες χώρες. Και αν ναι, υπό ποιους όρους. Πρέπει να υπάρχει η διαφάνεια, μήπως να υπάρχει απαγόρευση εξαγωγών. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μεγάλο αυτό το ζήτημα, δεν μας επηρεάζει ουσιαστικά το θέμα αυτό, φορά την Ασία και άλλο. Αλλά θεωρούμε ότι θα είναι ευκολότερο να βρεθεί μια μόνιμη λύση εάν ταυτοχρόνως ε, μπορούμε να δούμε αν υπάρξει μια ρύθμιση γενικότερη για αυτό το θέμα για να έχουν όλοι κάτι που θα αποκομίσουν από τη διάσκεψη την Υπουργική. Τρίτο θέμα, βαμβάκι, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες αυτές, Μαλή, Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο και Τσάντ, οι τέσσερις χώρες που εξαρτώνται από το Βαμβάκι. Υπάρχει εντολή του ΠΟΕ για να δούμε το θέμα πιο φιλόδοξα από ότι άλλους τομείς, δηλαδή για τις επιδοτήσεις και τους δασμούς. Υπάρχει μια πρόταση να καταργηθούν και τα δύο ταυτόχρονα, κάτι το οποίο δεν θα γίνει γιατί η Κίνα και η ΙΠΑ επιδοτούν την εγχώρια παραγωγή τους πολύ. Από τη σκοπιά της Ένωσης δεν έχουμε ε, κάτι στο πορτοκαλί κουτί για επιδοτήσεις ε, βάμβακα. Έχουμε όμως ένα περιορισμένο ποσοστό στήριξης για ε, τους Έλληνες και Ισπανούς παραγωγούς. Ήταν κομμάτι της συνθήκης ένταξης Ελλάδας και Ισπανίας και τους ε, στηρίζουμε με 270 εκατομμύρια ετησίως. Δεν είναι τραγικό ποσό όταν μιλάμε για γεωργική στήριξη, ε, αλλά δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε γιατί είναι στην συνθήκη ένταξης και το επίπεδο αυτό. Και ούτως ή άλλως η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με τις διεθνείς τιμές, ε, δεν τις καθορίζουμε εμείς. Και το τέταρτο θέμα, η πιθανή απαγόρευση ε, απαγόρευσης εξαγωγών, δηλαδή κάποιες χώρες όπως η Ινδία αλλά και η Ουκρανία, Ρωσία επιβάλλουν απαγόρευση εξαγωγών δημητριακών για λόγους διατροφικής ασφάλειας ή για να έχουν κάποιο πλέον έκτημα η παραγωγή τους. Οι απαγορεύσεις αυτές βεβαίως ε, ε, καταλήγουν να βλάπτουν, τους, ε, να βλάπτουν άλλες χώρες π.χ. την διατροφική του ασφάλεια, την πρόσβαση σε βασικά χαθά, κερδοσκοπία και κάποιες βεβιασμένες αγορές και δεν είναι κατωθετικό. θετικό. Κάποιες χώρες, ειδικά αυτές οι οποίες εξαρτώνται από τις εισαγωγέ για τα γεωργικά προϊόντα, έχουν ζητήσει νέους κανόνες του ΠΟΕ για να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτές τις απαγορεύσεις εξαγωγών. Δεν νομίζω να το καταφέρουμε. Αυτό το οποίο θα έχουμε μάλλον είναι περισσότερη διαφάνεια και κάποια προειδοποίηση. Είναι νομίζω σαφές από αυτά τα οποία είπα ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για τα αποτελέσματα του ΠΟΕ τον επόμενο μήνα. Οπότε, ποιε είναι οι προοπτικές. Εμείς είμαστε φίλοι του συστήματος αυτού, θέλουμε να ενισχύσουμε τους κανόνε αλλά δεν θέλουμε να γίνει αυτό με οποιοδήποτε τίμημα, ούτε να είμαστε εμείς οι μόνοι που πληρώνουμε. Θεωρούμε ότι έχουμε κάποιες ρεαλιστικές προτάσεις με σταδιακά βήματα και το ότι το καταφέραμε αυτό με τη Βραζιλία και με άλλες χώρες νομίζω καταδεικνύει ότι τώρα βρισκόμαστε κάπου στο κέντρο και δεν είμαστε σε αμυντική θέση αλλά δεν μπορούμε βεβαίως μόνοι μας να τα κινήσουμε την διαδικασία, χρειαζόμαστε και στήριξη και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια συνένεση για τις πρόπτικες ε, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις των που Οι ΙΠΑ δεν έχουν ε, όρεξη για περισσότερες ε, τέτοιες διαπραγματεύσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια αποφεύγουν τις πολυμερείς συνθήκες για τους λόγους που ξέρετε. Η Ινδία είναι σε αμυντική θέση. Η Κίνα έχει το δικό της πρόγραμμα και, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνθήκη αναγκαία αλλά όχι ικανή για αλλαγές στον ΠΟΕ. Χρειαζόμαστε και άλλες χώρες. Όπως είπα, εμείς ενδιαφέρομαστε κυρίως για μεταρρυθμίση των εσωτερικών αυτών ενισχύσεων. Ε, δεν έχουμε πολύ σκληρή για το βαμβάκι και Γι' αυτά θα παλέψουν άλλες χώρες. Εάν δεν έχουμε κάποια πρόοδο στα ζητήματα που ανέφερα, αυτό το οποίο θα προκύψει ε, θα είναι απλά ένα πρόγραμμα εργασίας ε, για να προχωρήσουμε παραπέρα τα επόμενα δύο χρόνια στις προοπτικές περαιτέρω μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τις εσωτερικές ενισχύσεις. Αυτά από εμένα. Ε, θα εκπροσωπηθεί η γενική μας διεύθυνση και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ε, και βεβαίω αναμένουμε τη συνεργασία της αντιπροσωπείας μας με την προσωπία του Κοινοβουλίου στον Buenos Aires ε, και βεβαίω θα, θα είστε ενήμεροι για να υπάρχει μια ε, ενιαία παρουσία της Ένωσης και βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Είναι όντως πολύ σημαντικό να είμαστε σπηρωμένοι και να περιορίσουμε τις παραχωρήσεις και τη, την τις υποχωρήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με αυτά που είπατε. Πέραμε στη συζήτηση. Ο κύριος Αντρία είναι ο πρώτος. Αντρία είπαμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως τα σοφά λόγια που είπατε είναι πολύ επίκαιρα του Πρόεδρου εννοώ τόσο σοφαλόγια. Και σε μια στιγμή μάλιστα που όπως είπατε και εσείς, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, διαστόματο του Προέδρου του είναι στα πρόθυρα να, τον, να εγκαταλείψουν το ΠΟΕ. Σχεδόν το έχουν δηλώσει. Οπότε εμεί θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη σύνεση και σοφροσύνη στον Buenos Aires και λίγους μήνες ε, πριν τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, για το μέλλον της ΚΑΠ. Δεν πρέπει εμείς να είμαστε ε, ακριβώς επειδή είμαστε καλοί μαθητές στον ΠΟΕ να πάμε πολύ γρήγορα και πολύ μακριά και για τη δημόσια αποθεματοποίηση όταν βλέπουμε τι κάνουν οι υπόλοιπες ε, ήπειροι και χώρες καλό είναι να είμαστε οι πρώτοι μαθητές αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιποι να μας ακολουθούν δεν αρκεί να είμαστε ηγέτες θα πρέπει να έχουμε και κάποιους συμμάχους και για το Μερκοσούρ ε, είπαμε και το συζητήσαμε με τις Γενικές Διευθύνσεις Εμπορίου και Γεωργίας, είναι αδιανόητη συζήτηση το διαπραγματεύσεων με τη Μερκοσούρ χωρίς το κεφάλαιο εθανόλη και βόλιο κρέας. Και δεν θα πρέπει να ε, είναι η Γεωργία το θύμα της συμφωνίας αυτής. Και διαρωτόμαστε κατά πόσο έχουμε προχωρήσει σε αυτές τις συζητήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επαγρύπνηση, σε εγρήγορση για το μπλε κουτί που αναφέρατε, θα πρέπει και εκεί να είμαστε προσεκτικοί και να μην φτάσουμε πολύ γρήγορα σε ανώτατο όριο στο μπλε κουτί, όπως είπατε, γιατί θα μπορούσε το μπλε κουτί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να στηρίξουμε τους κλάδους μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ε, είπαμε ότι υπάρχουν κάποια ευαίσθητοι κλάδοι στη συμφωνία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στη συζήτηση του Buenos Aires. Ε, θα ήθελα να απευθύνω λοιπόν μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι επιφυλακτική και προσεκτική και σε εγρήγορση. Γιατί αν έχουμε αποτυχία της πολυμέρειας, παρόλο που υπάρχει ένα παράδοξο εδώ με τη δράση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά διμερών συμφωνιών και έχουμε μια, ένα παράδοξο μεταξύ της πρόθεσης της δηλωμένης υπέρ της πολυμέρειας και της δράσης ε, που επικεντρώνεται σε διμερείς συμφωνίες. Αυτά λοιπόν όλα θα πρέπει να τα σταθμίσουμε εν ώψη και της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ο κύριος Γιάρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρώτη καλή είδηση εδώ και χρόνια. Από την εποχή που ξεκίνησα να υπερασπίζομαι τις συμφωνίες ε, και στην εκλογική μου περιφέρεια Πάντα υποστήριζα ότι έπρεπε να, να ε, ενισχυθούν οι πολυμερείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες μέσω του ΠΟΕ. Πολύ καλό λοιπόν που ξαναρχίζουμε. Βεβαίως έχουν διατυπωθεί πολλές επικρίσεις από τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις. Έχει κάνει παραχωρήσεις πρώιμες η Γεωργία χωρίς ανταπόδοση και το σύστημά μας βλέπουμε ότι δεν μπόρεσε να εξαντλήσει ε, τους, τα, περιθώρια που είχε μέσα από το Yellow Box. Αυτό θα ήταν πολύ καλό βεβαίως με δεδομένο τώρα θα μειωθεί το Yellow Box, αλλά το λέω για να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί για τα περαιτέρω. Και η τελευταία μεγάλη μεταρρύθμιση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν ήταν ε, ανέμακτη, είχε, απέτησε πολλές θυσίε. Λοιπόν, έχουμε την ε, αποσύζευξη των ε, ενισχύσεων, πολύ καλά. Ωστόσο, το κομμάτι αυτό, το οποίο παραμένει στο yellow box ή πάει στο green box, στο πράσινο κουτί, το επισημαίνω διότι είχαμε πολλές συζητήσεις στη Γερμανία για το εάν υπάρχει δυνατότητα της σύζευξης ή όχι. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι μήπως είμαστε υπερβολικά γενναιόδοροι και μειώνουμε το τερότατο επίπεδο και αφήνουμε το Yellow Box σε ένα, ε, το κίτρινο κουτί σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα μας επιτρέπει στο μέλλον καμία αλλαγή. Πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη που λίγο πολύ έχει καλυφθεί η δημόσια αποθεματοποίηση δεν θα απαγορευτεί εν τέλει από την παγκόσμια αγορά. Εάν μια χώρα όπως η Ινδία αναπτύσσει μέσα από το σύστημα το τελωνιακό της ε, μια δημόσια αποθεματοποίηση ε, δεν θα πρέπει εμείς να το επισημάνουμε και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε από τη δική μας την πλευρά. Αυτά είναι σοβαρέ επιφυλάξει. Βεβαίω, πάντα λέμε ότι είναι πολύ θετικό το ότι ξαναγυρνούμε στι πολυμερεί διαπραγματεύσει στον ΠΟΕ, αλλά πρέπει και οι λύσει για τη γεωργία να είναι οι σωστέ. Πάντω χαίρομαι γιατί η πρόοδο η δική μα από τη δική μα πλευρά είναι τέτοια που δείχνει ότι δεν ισχύουν οι κατηγορίε που είχαμε στο παρελθόν ότι η γεωργία ήταν εκείνη που παρεμπόδιζε κάθε περαιτέρω πρόοδο στον ΠΟΕΤ. Τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να είναι και μοχλός υποστήριξης των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ κύριο Στάκουλα. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση που μας έκανε. Είναι σχεδόν σαφές ότι στην η επερχόμενη υπουργική διάσκεψη ενδέκατη θα είναι αρκετά δύσκολη και απαιτητική γιατί κάποια κρατημέλη δεν είναι τόσο ε, ενθουσιώδη με το Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οπότε καλό είναι να έχουμε φιλόδοξη ε, ατζέντα στο Buenos Aires και χαίρομαι που κρατούμε την ηγετική μας θέση σε αυτή τη συζήτηση. Η γεωργία είναι ένα από τα λίγα θέματα που έχουμε μεγάλες πιθανότητες για αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο επίκεντρο των συζητήσεων και υψηλή προτεραιότητα των συζητήσεων τη γεωργία. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών και να τι ενθαρρύνουμε να προσυπογράψουν και να εφαρμόσουν τους κοινού κανόνες, ιδιαίτερα στο θέμα της δημόσιας αποθεματοποίηση που μας ενδιαφέρει σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να ρωτήσω τρία πράγματα σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή την Αφρική στις συζητήσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ε, ποια είναι η θέση και η σχέση της Αφρικής με τη Γεωργία. Ε, αναφέρεται το θέμα της δημόσιας αποθεματοποίησης και στην Αφρική. Έχουμε κάποια νέα για το πώς θα επηρεάσει το Brexit τη Γεωργία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αυτά ευχαριστώ. Κύριο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ε, περιεκτική επισκόπηση που μας κάνατε. Ε, ε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα καθεστώς ε, επέμβαση στις συνδίκες κυβέρνησης ό,τι αφορά τη δημόσια αποθεματοποίηση. Σε ποια καλλιέργεια αναφέρεται αυτή η δημόσια αποθεματοποίηση, σε μία ή περισσότερες και αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται και οι αγορές παρεμβατικές ε, μετά δρομολογούνται στις εξαγωγές και άρα σε χαμηλές ε, τιμές, σε τιμές dumping. Γιατί δεν μπορούν πια να τις αποθεματοποιήσουν, να τις αποθηκεύσουν αυτές τις καλλιέργειες. Επίσης με εκνευρίζει κάπως ε, η άρνηση και μάλιστα εδώ στην Ολομέλεια. Πολύ συχνά αρνούμαστε να εγκρίνουμε κάποιες ποικιλίε ε, του και σόγιας επειδή είναι γενετικά τροποποιημένες και μάλιστα με επιχειρήματα που δεν έχουν σχέση με την ασφάλεια αλλά λόγω της ε, σταυροφορίας των οικολόγων, των πρασίνων. ποια είναι η θέση των υπόλοιπων χωρών για τα θέματα αυτά. Η κυρία Ράνς Γκαρσία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε, παρόλο που ε, μου έμειναν δύο σημαντικές ανησυχίες. Μιλήσατε για το περιορισμό του περιθωρίου του πορτοκαλί κουτιού. Πώς θα επηρεάσει ένα τέτοιο περιορισμό του περιθωρίου τα κράτη-μέλη, γιατί δεν χρησιμοποιούν όλοι με τον ίδιο τρόπο το πορτοκαλί κουτί και τις ενισχύσεις που μπορούν να χορηγούν. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό το θέμα τις υπόλοιπες 27 χώρες μέλη. Δεύτερη ανησυχία και προβληματισμός μου αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση του Τραμπ η πλειοψηφία τουλάχιστον υποχώρησε από το TTIP μια σημαντική πολύ για μας συμφωνία και αποχωρώντας από την θέση αυτή και μάλιστα με την αναγγελία ότι θα απο, απομακρυνθεί και από το παγκόσμιο εμπόριο δημιουργεί φοβέρε ανησυχίες. Επίσης έχουμε πρόβλημα με τις ε, ισπανικές εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών. Ε, φαίνεται ότι με πρόσχημα αυτό το προϊόν θέλει να αμφισβητήσει τις ε, ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις στη Γεωργία, οι Ηνωμένες Τη Ευρωπαϊκή Γεωργία. Πώ θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα. Δεν μα ενδιαφέρει τόσο το θέμα των επιτραπέζων έργων της Ισπανίας, αλλά το ότι αμφισβητείται η ανάγκη των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων στη Γεωργία από τις ΗΠΑ. Σα ευχαριστώ. Κύριο φλανναγκαν Σα ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, όπως πάντα κύριε Κλάρκ. Έχουμε στον πίνακα που βλέπουμε και η ερώτηση είναι το να είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρώτος μαθητής έχει κάποια ωφέλη. Γιατί όταν έχουμε ένα όριο που δεν το αξιοποιούμε και μάλιστα μια στιγμή που χρειάζονται στήριξη η γεωργία. Δεν ξέρω, είμαι περίεργος. Ποιο είναι το όφελος του να είμαστε οι καλύτεροι και να έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις, να είμαστε ο καλύτερος, ο πρώτος μαθητής στον ΠΟΕ. Επίσης, τι γνώμη έχετε από τις συνέπειες που θα έχει η παρουσία του πρόεδρου Τραμπ στις διαπραγματεύσεις. Ο κύριος Δάντα Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Κλάρκ. Μας, μας παρουσιάσατε τι μπορούμε να αποφύγουμε αλλά δεν μας παρουσιάσετε τι μπορούμε να κερδίσουμε από μια νέα συμφωνία στον ΠΟΕ. Γιατί καλό είναι να είναι κανείς αμυντικός, αλλά σε μια συμφωνία θέλουμε αμοιβαία ωφέλη. Τι μπορούμε εμείς να κερδίσουμε με αυτό το νέο γύρο της συζητήσεων στον ΠΟΕ, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε μελέτη επιπτώσεων από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ ψηλότερο κόστος παραγωγής, γιατί το βιωτικό μας επίπεδο είναι υψηλότερο από το επίπεδο των υπόλοιπων υπήρων, κάτι που δικαιολογεί το υψηλό επίπεδο επιδοτήσεων στην ΚΑΠ. Και σίγουρα στις αιτήσει έχουμε κάποια όπλα. Μειώνουμε τώρα το περιθώριο ελιγμών, αλλά η πραγματικότητα του μέσου κατακεφαλήν εισοδήματος στην Ευρώπη υπάρχει. Και το να στερούμαστε το περιθώριο ελιγμών μας είναι πολύ επικίνδυνο για τους επόμενους, για τους διαδόχους μας. Επίσης, το θέμα των παγκόσμιων αποθεμάτων. Νομίζω ότι αν αν περιμένουμε κάποια πρόοδο, είναι περισσότερη διαφάνεια στο θέμα των παγκόσμιων αποθεμάτων. Η ΦΑΟ, μετά το αίτημα το G20, έκανε μια μελέτη για την καταπολέμηση της αστάθειας των τιμών και τη διαχείριση των παγκοσμίων αποθεμάτων. Αν λοιπόν ο ΠΟΕ συμπεριλάβει στο διεντολογικό του κώδικα και αυτή τη μελέτη της ΦΑΟ, θα έχουμε σημειώσει ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα σημαντική πρόοδο για ένα ζήτημα που μας ταλανίζει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, τη φοβερή αστάθεια και μεγάλη διακύμανση των παγκοσμίων τιμών. Ευχαριστώ κύριο Νίκολσον. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Κλάρκ για την παρουσίαση που μας έκανε. Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλη την παρουσίαση γιατί ήμουν σε άλλη επιτροπή. Πάντως, ε, γνωρίζοντας τον κύριο Κλάρκ εδώ και πολλά χρόνια βλέπω ότι δεν είναι και πολύ αισιόδοξο και φυσικά έχει βάσιμου λόγου από την πείρα του που δεν δικαιολογούν υπερβολική αισιοδοξία. Τώρα, ε, τη στιγμή που ασχολούμαστε με, τα, με τις πολυμερείς πτυχές ε, του ΠΟΕΝΟ, ταυτόχρονα έχουμε διμερείς συζητήσεις. Ε, το είπε και ο κύριος Αντρία Οπότε έχουμε ένα παράδοξο και μη διαφορά και όλα αυτά δρομολογούνται ταυτόχρονα. Έχω λοιπόν μία ερώτηση. Είπατε, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε την επόμενη διετία. Οπότε μία διετία είναι μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα έχουμε καν δει το τέλος των συζητήσεων. Μία δική μου πάντως απορία είναι μήπως θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια συνολική συμφωνία παρά να έχουμε αυτές τις ε, επιμέρους διμερείς συμφωνίες που ανακύπτουν παράλληλα. Επίσης, ποιος είναι ο κίνδυνος. Γιατί ασχολούμαι με τον ΠΟ εδώ και πολλά χρόνια και πολλοί είναι επιποδός και προβληματίζονται και ανησυχούν. Αλλά αν δεν είχαμε τη συμφωνία του ΠΟΕ ε, εδώ και τόσα χρόνια δεν θα ήμασταν καλύτερα σήμερα από ότι με αυτέ τι μεμονωμένε συμφωνίε που γίνονται συνεχώ ή τι διμερεί. Θα ήταν καλύτερα αν είχαμε από παλιά μια παγκόσμια συμφωνία σε επίπεδο ΠΟΕ, γιατί οι επιμέρου συμφωνίε δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και δυσκολίε. Επίση, η κατάσταση στι Ηνωμένε Πολιτείε. Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και τη δέσμευση του Τραμπ υπέρ του πρώτα η Αμερική. Αυτό τουλάχιστον έλεγε αρχικά. Πριν από λίγες εβδομάδες ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και μου είπαν ρητά ότι δεν έχουν ε, καταργήσει ακόμη το TTIP. Ε, ότι πολύ ευχαρίστως θα ξαναλάβω μέρος σε συζητήσεις για το TTIP. Δεν το έχουν ξεγράψει τελείως. Οπότε υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις δεν θα ήταν λοιπόν καλύτερα να έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία από ενιαία να μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα από τις επιμέρους συμφωνίες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να απαντήσετε. Αλλά θα πρέπει να προβληματιστούμε και από άλλα θέματα, γιατί όλα τα προβλήματα που έχουμε δεν πρόκειται να εξαφανιστούν ούτε να διευκολυνθούν, μάλλον θα επιδεινωθούν. Δεν θα ήταν μήπως καλύτερο να ανασκουμποθούμε και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Ολοκληρώσαμε τις ε, ερωτήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Όπως είπε ο κύριος Νίκολσον, φαίνεται ότι το TTIP δεν έχει φύγει τελείως από τον ορίζοντα αλλά ίσως πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση. Τι είπα από τη μια ΠΟΕ, από την άλλη, δηλαδή διμερής διαπραγμάτευση, πολυμερής διαπραγμάτευση, πως υπάρχει ανταγωνισμός και τι είναι το καλύτερο τελικά, πολυμερής συμφωνίες ή διμερής, παρακαλώ. Κύριε Νίκολσον, λέτε ότι έρχομαι και σα περιγράφω ζωφερές εικόνες. Ο κύριος Φλάναγκαν μου λέει ότι παρά είμαι αισιόδοξο. Ε, για το πρώτο λοιπόν, το κύριο. Βεβαίω οι πολυμερείς λύσεις είναι καλύτερες από τις ημερείς. Το αντιλαμβανόμαι, θα πιστεύω όλοι. Γιατί έτσι και όλοι συμβάλλουν και όλοι υποφελούνται και πιο δίκαιες είναι αυτές. Αλλά στη τελευταία προσπάθεια πέσαμε με φόρα πάνω στον τοίχο γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα για πολυμερείς συμφωνίες και αναγκαστήκαμε και εμείς και άλλοι να περάσουμε στις διμερείς λύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για την πρόσβαση στην αγορά, για την κατάργηση των ε, δασμολογικών φραγμών, οι λύσει πλέον είναι μόνο διμερείς και προοπτική, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εγώ, στο προσεχές μέλλον από τον ΠΟΕ να δούμε νέο γύρο απελευθέρωση των δασμολογικών ε, φραγμών δεν μπορούμε να περιμένουμε. Παρόλα αυτά, κανόνες για επιδοτήσεις διμερώς δεν μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης μόνο πολυμερώς. Και γι' αυτό και μπορέσαμε πριν από δύο χρόνια στον ΠΟΕ να εξασφαλίσουμε την απάλληψη των εξαγωγικών, εξαγωγικών ενισχύσεων. Πολυμερό μόνο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και όχι διμερό. Και γι' αυτό τώρα προσπαθούμε να προβούμε και στο επόμενο βήμα, δηλαδή να ασκήσουμε την πίεση για να μειωθούν οι ε, χώριες ενισχύσεις που έχουν στρεβλωτικό για το εμπόριο χαρακτήρα. Πάλι πολυμερός μπορεί να επιτευχθεί αυτό και όχι διμερός. Αυτό δεν είναι θέμα επιλογής μεταξύ ε, συμφωνιών για εμπορικές συναλλαγές ή ΠΟΕ αφετέρου. Οι FTA έχουν να κάνουν με τους δεσμολογικούς περιορισμούς, ενώ στις εξαγωγές ενισχύσεις, ε, εξαγωγικές ενισχύσεις, ο ΠΟΕ είναι ο χώρος ο κατάλληλος για την επίτευξη των συμφωνιών που θέλουν αναγκαστικά πολυμερείς. Τώρα για τις άλλες παρατηρήσεις βεβαίως και συμμερίζομαι 100% της ε, προεδοποίησης του κύριου Άντριου, ε, βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον ΠΟΕ. Δεν είναι δυνατόν μονομερός εμείς να μειώσουμε τις δαπάνες μας από το κίτρινο κουτί. Πρέπει και οι άλλοι να προβούν σε αντίστοιχους περιορισμούς. Και βεβαίως εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τους, ε, τα παπαδοπαίδια και να προχωρήσουμε μονομερός σε κινήσεις καλής θελήσεως, πρέπει όλοι ταυτόχρονα να κινηθούν. Και όπως είπα, η αδίποτε λύση σχετική με τις εγχώριες ενισχύσεις θα ε, συναυθεί μόνο όταν δούμε ότι υπάρχει επαρκές περιθώριο για να συνεχίσουμε την πολιτική στήριξη είτε με την υπολοιπόμενη στήριξη που μπορούμε να έχουμε στο κίτρινο κουτί, είτε από το μπλε κουτί, είτε από το πράσινο κουτί. Και όταν μιλήσατε, κύριε Γιάρ, εσείς, για, το, για τις ενισχύσεις, είναι αυτό που ονομάζουμε ε, ενισχύσεις από το μπλε κουτί. Αυτές δηλαδή οι οποίες ε, δεν αυξάνουν την παραγωγή ή τις τιμές, αλλά στηρίζονται σε, ένα σε μια συγκεκριμένη έκταση εκτάρια ή αριθμό κεφαλιών, δηλαδή συγκεκριμένο ζωικό κεφάλαιο. Και εδώ η κίνησή μας είναι από τις τρευλωτικές του εμπορίου ενισχύσεις να περάσουμε στις ενισχύσεις του πράσινου κουτιού που είναι σύμφωνες με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και το πρασίνισμα. Αυτό μας ενδιαφέρει και κάθε διαπραγματεύση στο μέλλον για την ενίσχυση του μπλε κουτιού θα σημαίνει μια σταδιακή απάλληψη αυτών των ενισχύσεων του μπλε κουτιού με την ε, παράλληλη και τις μεταρρύθμισεις ε, της ΚΑΠ. Νομίζω, κύριε Ανδρίου, απάντησα στην ερώτηση για τις διμερείς ε, συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και τον ΠΟΕ. Στον ΠΟΕ έχουμε μόνο επιδοτήσεις ως θέμα συζητήσεων για τη δημόσια αποθεματοποίηση που ρώτησε ο κύριος Γιάρα αλλά και άλλοι. Το θέμα είναι ότι, όπως άλλωστε και εσείς είπατε, η Ινδία αγοράζει σε πολύ υψηλή τιμή από τους γεωργούς σίτο και όριζα, τα αποθεματοποιεί και τα πολύ σε πολύ χαμηλότερη τιμή, άρα ε, με τον τρόπο αυτό επιδοτεί τους παραγωγούς της και κάποιες από τις εξαγωγές αυτές, κάποια από ε, τις προσότητες αυτές πάνε στην εξαγωγή, έμεσα τουλάχιστον, ενώ χώρες όπως το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες που έχουν αντίστοιχη παραγωγή όριζας και σύτου, ε, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και για τη δυνατότητα του να πουλήσουν αγορά της Ινδίας και για τη δυνατότητά τους για εξαγωγές σε άλλες περιοχές της Ασίας. Αυτή είναι κατ' ουσίαν ε, η... Αυτές είναι οι δυσμενείς συνέπειες των δημόσιων, ε, της δημόσιας αποθεματοποίησης που μπορεί να έχει ρόλο προστατευτικό αλλά συνήθως ε, γίνεται κατάχρησή της για την παροχή έμεσων ενισχύσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα. Ρύζι και σιτάρι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Κάποιος βουλευτής επίσης είχε ρωτήσει για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και το κατά πόσον αποτελεί ε, σημείο τριβής με τις ΗΠΑ πολιτική για την ε, μη αποδοχή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στον ΠΟΕ, όχι, θα έλεγα, μπορεί να μην σα ικανοποιήσει αυτή η επιλογή, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει δεκτά περί τα 50 ε, στελέχη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, κυρίως ε, φασόλων, φασολίων ε, σόγιας, φασιόλων σόγιας, ε, κυρίως για ζωοτροφές, με μια διαδικασία η οποία τώρα προχωρεί ταχύτερα από ό,τι πριν. Οι ΔΕΗ Ηνωμένε έχουν αντιληφθεί ότι έχουμε τις σοβαρές μας επιφυλάξεις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Απλώς επισημαίνουν ότι δεν γινόταν, επισήμαναν μάλλον, επισήμεναν ότι δεν γινόταν αρκετά γρήγορα η εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων, των ισιών των κανόνων. Ενώ τώρα και αυτό έχει αντιμετωπιστεί γιατί προχωρεί επρόσκοπτα η διαδικασία και δεν βλέπω να διατυπώνονται ενστάσεις ή επιφυλάξεις από τις ΗΠΑ για τα ους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ο κύριος Τάκουλα ρώτησε τι λένε οι αφρικανικές χώρες για τα θέματα που σας επισήμανα. Κοιτάξτε, οι αφρικανικές χώρες δεν έχουν μία Στάσει στην υπόθεση αυτή. Είναι αρκετά διαφορετικέ οι θέσει του ανάλογα με την οικονομική και την πολιτική κατάσταση που γνωρίζει κάθε χώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται δηλαδή για μια ενιαία ομάδα κρατών με κίνηση προ την ίδια κατεύθυνση πάντα. Αλλά πάντω. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν θέλουν να τους ε, απορροφήσουν κάποιες συμφωνίες που θα ληφθούν και πάνω απ' όλα όχι αυτές που έχουν να κάνουν με αναπτυσσόμενες χώρες. Και βέβαια εδώ ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι απαραίτητα αυτές οι οποίες προξενούν στρεβλό στην αγορά των γεωργικών προϊόντων. Η Κίνα και η Ινδία επιτοπλίστων που ξοδεύουν πολύ δημόσιο χρήμα στρεβλώντας έτσι την αγορά και ως εκ τούτου τις ε, δυνατότητες που έχουν ε, να διαθέσουν την παραγωγή τους οι αφρικανικές χώρες. Στον Βάμβακα, παραδείγματι, των δυτικοαφρικανικών κρατών το πρόβλημα δεν έγκυται στην υποστήριξη μπορεί να δίνει, στην ενίσχυση μπορεί να δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο βάμβακα τη Ισπανία ή τη Ελλάδα, στα γόνα στον ωκεανό αυτό. Αλλά αντίθετα, στι κινήσει τη κίνα που ε, επιδοτούν το βαμβάκι του για να γίνει πολύ ανταγωνιστικό στον κόσμο και έτσι πλήττουν αυτέ τι πολύ πιο φτωχέ αναπτυσσόμενε χώρε. Στο Brexit θα περάσω στο τέλο ε, τη τοποθέτησή μου για την κυρία Εράντς Καρσία. Ε, γύρατε πολύ εύστοχες παρατηρήσεις ίσως να μην το τόνισα αρκετά, επιτρέψτε μου να επανέλθω και να το τονίσω, να το επαναλάβω, δεν πρόκειται να δεχθούμε νέους κανόνες για τη γεωργία από τον ΠΟΕ, κανόνες δηλαδή που θα μας απαγόρευαν τη χρήση ή την αξιοποίηση του περιθωρίου που έχουμε για ενισχύσει μέσω του κίτρινου του μπλε κουτιού ή που θα περιορίζαν τη δυνατότητά μας στο μέλλον ε, αν δηλαδή θέλουν τα μέλη του ΠΟΕ να προβούν όπως και εμείς σε μεταρρυθμίσεις, πολύ ευχαριστώ. Αλλά μεταρρυθμίσεις μόνοι μας δεν πρόκειται να κάνουμε, δεν θα περιορίσουμε δηλαδή το περιθώριο χειρισμών μας ε, μέσα από αυτό. Αναφερθήκατε σε μια σειρά από συγκεκριμένε υποθέσεις, περιπτώσεις και ανησυχίε σχετικές με τις ΗΠΑ, ημιλήματα. Φανταζόμαι ότι θα μιλούσατε για τις ε, ελιές ότι δεν θα μιλούσατε για τις ελιές, μιλήσατε όμως. Ναι, όντως υπάρχουν μια σειρά από φραγμοί εμπορική σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η δυνάμη φραγμή. Ε, επεξεργαζόμαστε διάφορες λύσεις ε, για να μπορέσουμε να ε, γλιτώσουμε από τα προβλήματα αυτά. Ο κύριος Δεκάστρο και η Λυπή βεβαίως όταν επισκεφθούν τη Ουάσιγκτον το Δεκέμβριο στο πλαίσιο της ομάδας για τις διατλαντικές σχέσεις φαντάζομαι και θα παρακολουθώ βέβαια την, ε, την, ε, τις εξελίξεις και ό,τι θα έχουν να μας μεταφέρουν στη συνέχεια θα μεταφέρουν αυτές τις ανησυχίες των, το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε πρόκειται για το Ισελιέ είτε πρόκειται για τον Νίνο ε, ή για άλλα προϊόντα. Κύριε Φλάναγκαν, εσείς ρωτήσατε τι συνέπειες φέρνει για τον ΠΟΕ η ανάδειξη στην Προεδρία των ΗΠΑ του Τραμπ δεν ενδιαφέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες ε, ε, δεν ενδιαφέρονται οι ΗΠΑ για διαπραγμάτευση πολυμερών συμφωνιών αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό έχει φέρει. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή εστιάζονται στο σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, στο οποίο αποδίδουν ε, μια υπερβολική δικαστική δυνατότητα παρέμβασης αρμοδιότητες υπερβολικές και αυτές θέλουν να περικόψουν. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή βεβαίως μπορούμε ε, εμείς να προχωρήσουμε σε συμφωνίες σημαντικές στον ΠΟΕ χωρίς τις ΗΠΑ ελπίζουμε ότι η στάση τους θα αλλάξει στο μέλλον για τον κύριο Νίκολσον δεν είμαι σίγουρος ότι ε, αντελήφθηνε το επιχείρημα σε σχέση με τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και ΠΟΕ και την αντιπαράθεση είναι επιλογή αυτό τόσο ή άλλως Λυπούμε που χάθηκε η ευκαιρία μέσα από τον ΠΟΕ ε, για πολυμερει συμφωνίες. Ε, συμφωνώ, χάθηκε μια σπουδαία ε, ευκαιρία, αλλά η δεύτερη καλύτερη λύση, η επόμενη καλύτερη λύση είναι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Ο κύριος Τακούλα απεχώρησε δυστυχώς. Για τον Brexit όμως θα απαντήσω Ναι, ναι, και εσείς το είπατε κύριε Πρόεδρε. Για το Brexit λοιπόν ε, δεν βλέπω ότι θα φέρει μεγάλη διαφορά από το εξή. Δύο θέματα σχετικά με το Brexit ε, είναι σε κρεμότητα στον ΠΟΕ αυτή τη στιγμή. Η διαχείριση των ποσοστώσεων δασμολογικού χαρακτήρα με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και δεύτερον, πώς ή πότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει το χρονοδιάγραμμα για τις εθνικές του ενισχύσεις, ποιο θα είναι το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου και τι θα αντιστοιχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Εδώ λοιπόν, για να περάσουμε στο κίτρινο κουτί, στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα και που έχει να κάνει με την, ε, τις ενισχύσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιορίζονται από έναν το επίπεδο από μία οροφή, το χαμηλότερο κομμάτι δηλαδή στο γράφημα που βλέπετε στη γραφική παράσταση, το κίτρινο κουμπί με 110 δις αυτή τη στιγμή, από τα οποία η Ευρώπη των 28 δαπανά τα 9 ή 10 δις, εξαντλεί τα 9 ή 10 Από αυτά λοιπόν πώς θα υπολογιστεί το ποσοστό του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα κοιτάξουμε ποιο ήταν το ποσοστό του Ηνωμένου Βασιλείου όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν 12 τα κράτη-μέλη και αυτό θα είναι το ποσοστό του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση για τη μεθοδολογία αυτή. Γιατί στις περαιτέρω διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε ε, το περιθώριο του κίτρινου κουτιού και το ποσό που μπορούσε να δαπανίσει η Ευρώπη με τα νέα της κράτη-μέλη. Άρα μπορούμε να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή και αφαιρώντας τα πρόσθετα αυτά ποσά να φτάσουμε στο συνολικό, στον όγκο που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που εντάχθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο και με αυτό να υπολογίσουμε το ποσοστό που αντιστοιχεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Brexit. Επίσης, ένα ποσοστό ε, των ποσοστών δασμολογικού χαρακτήρα. Ας πούμε ότι έχουμε 110 τόνους ε, κράτος πουλερικών. Το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ορίσει ένα δικό του σχέδιο ή ε, κατάστοιχο ε, ποσοστό οντοσμολογικού χαρακτήρα για το κρέας πουλερικών. Άρα παίρνουμε τα 110 αυτά, τους 110.000 τόνους, βλέπουμε πόσο από αυτό το μερίδιο είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, ας πούμε ότι είναι 5.000 τόνοι, και άρα ή 15.000 καλύτερα. Οπότε το, στο μέλλον το TRQ αυτό, το ποσοστό δηλαδή των ε, ποσοστό συνδεσμολογικού χαρακτήρα για την Ευρώπη των 27 θα είναι 85.000 τόνοι, για το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι 15.000 τόνοι και αυτό πάλι με βάση τους, ε, τις μετρήσεις που είχαν γίνει με τις ε, διάφορες διευρύνσεις. Δηλαδή η ιστορία είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι είτε πρόκειται για διεύρυνση είτε πρόκειται για συστολή της ε, Δεσμολογικής Ένωσης της Θελωνιακής Ένωσης δεν επηρεάζονται οι λοιπές χώρες, οι τρίτες χώρες από την αύξηση στη μείωση του αριθμού των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα καταγραφεί και με το Brexit. Αντίστοιχα, για τη ζάχαρη, για το ε, πρόβιο κρέας, οποροκυπευτικά, ξέρετε ποια είναι η ύποπτοι, θα γίνει αντίστοιχη προσαρμογή και ο επιμερισμός αφενός της Ευρώπης, για την Ευρώπη των 27 και αφετέρου για το Ηνωμένο Βασίλειο. Χωρίς να υπάρχει ακόμα συμφωνία, ε, σε συζητήσει είμαστε ακόμα με τους εταίρους του ΠΟΕ. Πριν από τρεις εβδομάδες ε, κάναμε την παρουσίαση των προτάσεων στη Γενέβη. Βεβαίως η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εταίροι έχουν ερωτήσεις για να δευκρινιστεί αν είναι σωστές οι στατιστικές που τους παρουσιάζουμε και βεβαίως είμαστε πάντα πρόθυμοι να δώσουμε τις απαντήσεις και να προβούμε στις συζητήσεις που χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε κύριε Δευθυντά για τις διευκρινήσεις, τις απαντήσεις, την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Πιστεύουμε ότι θα είναι θετικό το αποτέλεσμα των συζητήσεων στον Buenos Aires. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και με πολύ μεγάλη χαρά θα σας ξαναπεριμένουμε στην Επιτροπή για την ενημέρωση της πρόοδου και των συζητήσεων από τον Buenos Aires. Ωραία, ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στις ε, συζητήσεις που θα γίνουν στον Buenos Aires. Ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, Γυρίζουμε τώρα πίσω στο σημείο 7 και ευχαριστώ θερμά την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Νταντσίλα, που συμφώνησε να συζητήσουμε πρώτα την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Νταντσίλα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της, που θέμα έχει τις μειονεκτούσες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για γνωμοδότηση επί της έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θέλουμε να τονίσουμε την σημαντική συμμετοχή που μπορεί να έχουν οι μενοκτούς περιοχές για την αναβίωση της υπαίθρου στο θέμα αυτό. κυρία η συγγήτρια έχει το λόγο παρακαλώ, κυρία Ντάντσιλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τις πιο πλούσιες περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν όμως ε, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ε, περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το εισόδημα ε, και τις ευκαιρίες. 47 από περιοχές από 8 χώρες μέλη θεωρούνται ε, περιοχές με χαμηλή ε, ανάπτυξη και με ΑΕΠ κάτω από 90% σε σχέση με το κοινοτικό μέσο όρο και μάλιστα χωρίς σταθερή ε, ανάπτυξη και χωρίς να έχουν επιτύχει ακόμη το αποθετό επίπεδο σύγκλησης. Επίσης έχουμε άλλες περιφέρειες με μια τάση αύξηση του ΑΕΠ κατά κεφαλήν, αλλά ακόμη δεν έχουν ξεπεράσει το 50% του κοινοτικού μέσου όρου. Έχουμε τέτοιες περιοχές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σε πολλές από τις περιοχές αυτές η γεωργία είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός παράγοντας και σημαντική πηγή εισοδήματο για τον πληθυσμό. Και γι' αυτό ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ αποτελεί κέρια σημασία χρηματοδοτικό μέσο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης ε, στην ύπεθρο των μειονεκτουσών περιοχών και ταυτόχρονα προσφέρει τα οικονομικά κίνητρα που απαιτούνται για να καλυφθούν οι συγκεκριμένες ε, εδαφικές ανάγκες αυτών των περιοχών. Η Γεωργία παρέχει ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό απασχόληση σε περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλει στην ε, δημιουργία υφόρου ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα το αναπτυξιακό με τις υπόλοιπες περιφέρειες και να διαφυλαχθεί η παραμονή του πληθυσμού στην Ήπεθρο. Ε, χρειάζονται όμως ε, ε, κονδύλια προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών αυτών με σχέδια που θα ξεκινούν από τη βάση προς τα πάνω. Και μάλιστα η συμμετοχή τοπικών ομάδων δράση στην ανάπτυξη των τοπικών στρατηγικών είναι ευπρόσδεκτη και για να στηρίξουμε τέτοια συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων ε, και να προωθήσουμε την αξιολόγηση και έγκριση μεμονωμένων έργων του Λίδερ χρειάζεται συνεργασία. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε ανάπτυξη υποδομών και ευρυζωνικές ε, συνδέσεις. Έτσι θα κρατήσουμε τον αγροτικό πληθυσμό στην Ήπεθρο και θα προσελκύσουμε τους απαραίτητους εργαζόμενους και μάλιστα ειδικευμένο εργατικό δυναμικό στις περιφέρειες αυτές. Χρειαζόμαστε καλή διασύνδεση των περιφερειών αυτών με το ψηφιακό δίκτυο, κάτι που θα αποτελέσει κίνητρο για συμπράξεις ερευνητικές και καινοτόμες, προκειμένου να βρεθούν καινοτόμε πρακτικές και να βοηθήσουν την εδραίωση και ανάπτυξη της γεωργίας και της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές ε, των πιο ε, μειονεκτουσών περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σε γενικές γραμμές λέω στη γνωμοδότησή μου και περιμένω τις προτάσεις και τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Σαντρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Βιόριτσα Νταντσίλα και να τη συγχαρώ για τη γνωμοδότησή της που είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι αρμόδια κατ' ουσία και αισθενίζομαι σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της γνωμοδότησης, ιδιαίτερα την ανάγκη Παγκόσμια στρατηγικής, ε, σφαιρικής, ε, συνολικής ανάπτυξης, ε, ιδιαίτερα των μειονεκτησών περιοχών. Αναφέρεστε στην πρωτοβουλία Leader, είναι πολύ σημαντική και ε, μιλάτε για την ανάγκη μιας προσέγγισης που θα ξεκινάει από τη βάση προς τα πάνω και την ε, συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης να αξιοποιήσουμε το σημαντικό δυναμικό και το αγροτικό, μεταξύ άλλων, στις μειονεκτούς περιοχές, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη επαρκώς. Γι' αυτό θέλουμε μια συνολική σφαιρική στρατηγική που θα βοηθήσει τις μειονεκτούς περιοχές να οργανωθούν καλύτερα, όπως το Πιεμόντε ή τις ορεινές περιοχές ε, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα μειονεκτήματα. Επίσης κάτι άλλο που είναι σημαντικό στη γνωμοδότηση και θα υποβάλλω και σχετικές τροπολογίες, ε, κάτι που αναφέρουμε πολύ αλλά δεν το οργανώνουμε, ε, τη σχέση μεταξύ αγροτικών περιοχών και αστικών περιοχών. Έχουμε σημαντικούς πόλους που θα πρέπει να εξορροπούνται μεταξύ τους και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στη μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινή γεωρικής πολιτικής και να βρούμε κάποιες γέφυρες μεταξύ των αστικών πόλων και των αγροτικών ζωνών. Αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα διακυβεύματα που θα μας βοηθήσει στην ανάπτυξη και της γεωργίας αλλά και της υπαίθρου μας στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Μίουλερ. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, του Χαντάκουλα θα μιλήσω, του Σκιώδους Συγητού. Και εμείς ε, βεβαίως σύμφωνο με την έκθεση της κυρίας ε, Τζαντσίλα, η οποία είναι ισορροπημένη και φοβόμαστε δυστυχώς ότι στο πλαίσιο του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου θα ασκηθεί πίεση στο Ταμείο Συνοχής Επίσης ε, θεωρούμε αναγκαίο να μην υπάρξει περιορισμός ε, των ε, περιοχών αυτών που έχουν μόνο χαμηλό σύνδημα, αλλά να ληφθεί υπόψη και η χαμηλή ανάπτυξη για εμάς είναι πολύ σημαντικό στο σημείο 2 να αναφερθεί και να τονιστεί ότι στο πλαίσιο των έργων leader θα πρέπει να δούμε αυτή την αρχή bottom-up και οι ομάδες δράσης να συνεισφέρουν πραγματικά. Το άλλο θέμα είναι η ψηφιοποίηση, το οποίο βεβαίως θέλουμε να το δούμε πιο στενά, γιατί μπορεί να είναι μια ευκαιρία βεβαίως, αλλά α, πιθανώς ε, να οδηγήσει κάπου και σε απώλειες ε, θέσεων εργασίας. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία και μια δυνατότητα εκπαίδευσης και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτές οι συνεργασίες για την καινοτομία. Ε, εδώ πάρα πολλές χώρες έχουν ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο, ειδικά αυτές ε, οι συνεργασίες που βασίζονται σε δικτύωση και βέλτιστες πρακτικές πραγματικά πρέπει να προωθηθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ροπέ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την κυρία Ταντσίλα. Είναι πολύ σημαντική η εκθέσή της. Ίσως περισσότερο για ορισμένα κράτη-μέλη από ότι κάποια άλλα, αλλά πάντως έχει τεράστια σημασία για τα πιο απομακρυσμένα κράτη, αυτή της περιφέρειας των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως αυτά που έχουν σύνορα κοινά με χώρες που έχουν ακόμη χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Είναι πολλοί οι λόγοι των αποκλήσεων στο βιωτικό επίπεδο μεταξύ υπαίθρου και αστικών κέντρων. Δεν έχουμε μπορέσει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ε, διαφορά, αυτά τα χάσματα. Και γιατί η παλαιά αλλά και η νεότερη γενναία τίνει, τίνουν να αποχωρούν από την Ήπεθρο και να συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι δεν βλέπουν σαφείς προοπτικές για το μέλλον. Ναι, μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχουν συστήματα υποστήριξη, αλλά στι προσεχεί δημοσιονομικέ προοπτικέ τι θα γίνει. Γνωρίζουν ε, οι άνθρωποι αυτοί τι θα συμβεί. Όχι, είναι σε μια κατάσταση εκκρεμότητα. Δεν γνωρίζουν τι θα φέρει το μέλλον για τις ε, περιοχές αυτές, τις οποίες φθήνει διαρκώς η γεωργική ε, δραστηριότητα και ιδιαίτερα στις ε, περιοχές όπου δεν μπορεί να είναι καθαρά προβλέψιμο ή ορατό το μέλλον, ή που μπορεί να είναι πιο υψηλός ο πληθωρισμός, να κρυβαίνουν πιο πολύ ε, οι συνθήκες παραγωγής, ε, ο κόσμος φεύγει, αποχωρεί από την Ήπεθρο για να συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα. Και βέβαια, Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε εδώ και καιρό, γιατί πρώτα κανείς ε, εστιάζεται, εγκαταλείπει την κτηνοτροφία που είναι πιο απαιτητική για να περάσει στην ε, φυτοκαλλιέργεια που έχει λιγότερες ε, δυσκολίες και μετά περνά, εγκαταλείπει τελείω την υπαίθρο και περνάει στην ε, πόλη. Άνισο λοιπόν βιωτικό επίπεδο. Επίσης άνισα και τα επίπεδα των ενισχύσεων μέχρι και κατά λόγο ένα προς ένα δεύτερο και υποτίθεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε ότι μπορούσε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έκανε ό,τι μπορούσε για να μειώσει αυτές τις αποκλήσεις, για να γίνει πιο ομοιόμορφη η Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο ελπίζω ότι θα επιτευχθεί σύν το χρόνο και με τις προσοχές προ... δημοσιονομικές προοπτικές θα έχουμε όλα τα ίδια επίπεδα ενισχύσεων και ε, βιωτικού επίπεδου και βιωτικά επίπεδα. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι η υποστήριξη από προγράμματα όπως το Leader που έχουν πολλές φορές πολύ περιορισμένη ε, πρικοδότηση ή είναι πολύ αυστηρά στην περιγραφή των προϋποθέσεών τους. Α τα κοιτάξουμε λοιπόν όλα αυτά. Α κοιτάξουμε αν υπάρχει δυνατότητα για συμπληρωματικά προγράμματα. Γιατί ο πυρήνα του Λίτερ έχει περιοριστεί πάρα πολύ και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήθελα παρακαλώ συλλαμβάνω το λόγο να μιλούν περισσότερο από ό,τι μίλησε η συντάκτρια τη γνωμοδότηση. Ο κύριο Φλάναγκαν. Καλή ιδέα, πρόεδρε, ναι, συμφωνώ. Έχουμε περιοχές οι οποίε εξαρτώνται περισσότερο από την χρηματοδότηση του πυλώνα 2, αλλά για απλοποίηση δεν γίνεται λόγος, ιδιαίτερα στο δεύτερο πυλώνα. Και έτσι η χρηματοδότηση, σε μεγάλο βαθμό η χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη, διατίθεται ε, μέσω ημικρατικών υπηρεσιών. Και ιδιαίτερα θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο για την έκθεση. Ένα πράγμα νομίζω μπορούν να κάνουν οι ευρωβουλευτές για να βοηθήσουν τις ε, περιοχές που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Και ξέρω ότι θα μου πει ο Πρόεδρος ότι δευτεριάτη κάτι τα λέμε όλα αυτά και όλα αυτά. Αλλά μπορούν να κάνουν κάτι οι ευρωβουλευτές. Είναι να πάνε να αρχίσουν να πιάσουν τη δουλειά στις περιοχές αυτές, να υπάρχει κόσμος που θα δουλέψει γιατί έχουν ε, απεριμωθεί τελείως. Ευχαριστώ, όντως, τι έχετε. Πολύ συχνά στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές ε, συνήθως όταν σκεφτόμαστε τις περιοχές ε, νομίζουμε ότι είναι οι απόμακρες ε, οι είναι νησιωτικές ή ορεινές, αλλά περισσότερες φορές και στην οδοχώρα, στο εσωτερικό των χωρών έχουμε τέτοιες περιφέρειες που υστερούν στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και το δεύτερο είναι ότι η πολιτική συνοχή αφιέρωσε κάποια κονδύλια στις περιοχές αυτές, στις περιφέρειες αυτές, αλλά όχι αρκετά κατά τη γνώμη μου. λίγα είναι τα κονδύλια της, Ευρω... της πολιτικής συνοχής που κατευθύνεται προς, τις, ε, προς την Ήπεθρο ή τις ε, μειονεκτούσες ή τις περιοχές που υστερούν στην ανάπτυξη, παρόλο που κοπτόμαστε υποτίθεται για την εδαφική συνοχή. Αυτά ευχαριστώ η τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα για τις περιφέρειες που υστερούν στην ανάπτυξη η γεωργία είναι ένας πολύ σημαντικός οικονομικός κλάδος και για πολλές περιοχές το πιο η πιο σημαντική πηγή εισοδήματος. Πάντως είμαι βεβαία ότι οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους θα εμπλουτίσουν τη γνωμοδότηση ε, και πραγματικά περιμένω τις τροπολογίες σας γιατί πραγματικά κάθε τροπολογία θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα συγκεκριμένης περιφέρειας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι τροπολογίες που θα καταθέσετε να ενταχθούν στην έκθεση και χάρη σε όλα αυτά να φανούμε πραγματικά χρήσιμοι για αυτές τις περιοχές που υστερούν στην ανάπτυξη. Περιμένω με ανυπομονησία τη ε, συνεισφορά σας και τις τροπολογίες. Μέχρι 10 Νοεμβρίου έχετε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τον Ιανουάριο θα έχουμε την ψηφοφορία και το τελευταίο θέμα είναι ο κανονισμός 1306, μάλιστα το σχετικό διορθωτικό για τον κανονισμό 1306 του 2013 και ε, από τη στιγμή που δεν έχουν υποβληθεί, όπως είπαμε, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ε, παρατηρήσεις ή εστάσεις ε, για, για το διορθωτικό αυτό, το δεχόμαστε και το παραπέμπουμε όπως πρέπει. Ραντεβού στις 9 την Πέμπτη θα έχουμε και ψηφοφορίες. Γι' αυτό μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Ευχαριστώ και τους διερμήνες, λέει ο Πρόεδρος, και κυρίως το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής ε, Γεωργίας.